Um, Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας. Έχουμε μια, ένα φορτωμένο πρόγραμμα μπροστά μας. Οπότε ας μην ε, χρονοτριβούμε. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ξεκινούμε από την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχει έτοιμο από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες να αναβληθεί το σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Οι ψηφοφορίες η διμερής ρήτρα διασφάλισης της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Κορέας. Οπότε, αντί για το σημείο 5 σήμερα, θα συζητήσουμε το σημείο 20, τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών αυτή καθεαυτή με την Κορέα. Οπότε θα αναλάβει και ο εισηγητής μας ο κύριος Στέρντι. Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτή την αλλαγή. Mm. Οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έχουμε επίσης τα πρακτικά της συνεδρίασης της 1 η Ιουνίου προς έγκριση. Τα θεωρούμε εγκεκριμένα αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Και τώρα οι ανακοινώσει Τι, την αλληλογραφία μας την έχετε στους φακέλους σας. Η συνάντησή μας θα περάσει και στο webstream του Κοινοβουλίου, εκτός βεβαίως από το μέρο τη συνεδρίας που ήταν και των θυρών. Και με αυτή την ευκαιρία να καλωσορίσω την κυρία, την κυρία Ελένα Χόλντορ Φρομέρο και τον κύριο Μπέντζαμιν Ρέι από τη δίκηση. Η κυρία Μωρέρα αντικαθιστά τον κύριο Σάπιν, ο οποίος έφυγε από την υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ουάσιγκτον και ο Μπέντζαμιν Ρέι αντικαθιστά τη Μερσέντες Ροντρίγκε, η οποία έχει άδεια μητρότητα για το ερχόμενο εξάμεινο. Καλώ ήρθατε λοιπόν και δυο σα. Να περάσουμε στο σημείο 4 εξέταση των τροπολογιών για το θέμα της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών και όπως αποφασίσαμε δεν θα ψηφίσουμε σήμερα αναβάλουμε την ψηφοφορία για αύριο όμως μπορούμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες δίνω λοιπόν το λόγο μάλλον όπως γνωρίζετε, υπήρξε ένα νομικό θέμα εδώ, ένα νομικό ζήτημα σε ό,τι αφορά το κατά πόσο είναι δυνατό ή όχι από νομική άποψη να υπάρχει περιφερειακή ρήτρα διασφάλιση. Ζητήσαμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Οπότε Διερωτώ με αν ο κύριος Πάσελς είναι μαζί μας. Όχι, ακόμη. still there is... Όχι, υπάρχει κάποιος από την νομική υπηρεσία ούτως ή άλλως. Η κυρία Γκάουτσι, η κυρία Γκάουτσι θα μας ανακοινώσει την άποψη της ε, νομικής υπηρεσίας για το θέμα της περιφερειακής ρήτρας Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα ζητήθηκε να εξετάσουμε κατά πόσον η περιφερειακή ρήτρα είναι νομικώς βιώσιμη ή όχι. Κατά πρώτον, πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία θεωρεί ότι η ρήτρα αυτή ισχύει για την τοπική βιομηχανία, αλλά δεν την καθορίζει. Η Επιτροπή επιχειρεί ένα ορισμό στην πρότασή τη, λέγοντας αναφέρεται μάλλον στους παραγωγούς της Ένωσης συνολικά των παρομοίων ανταγωνιστικών προϊόντων της Ένωσης ή τους παραγωγούς της Ένωσης που η συνολική παραγωγή τους των παρόμοιων ή των ίδιων ανταγωνιστικών προϊόντων θεωρούνται αναλογία της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής αυτών των προϊόντων. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν μπορεί να ενεργοποιηθεί μια ρήτρα εάν οι προποθέσει αυτέ δεν ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά σε μια περισσότερε περιφέρειε, περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από νομική άποψη, όταν εφαρμόζουμε μια διεθνή συμφωνία, πρέπει ω θεσμικά όργανα να διασφαλίζουμε ότι δεν προβλέπουμε μέτρα, αντικείμενα προς την ε, ουσία της συμφωνίας κατά πρώτον. Και έπειτα, ακόμη πιο σημαντικό, ότι δεν προβλέπουν μέτρα που υποβαθμίζουν τα δικαιώματα που έχουν προκύψει για το τρίτο μέρος μέσα από τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με την Κορέα ε, και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, αντιμετωπίστηκε ως μία ενιαία αγορά. Ήταν συνολική δηλαδή η εξέταση της ευρωπαϊκής αγοράς και το ίδιο και για την δημοκρατία της Κορέας. Ωστόσο, εφόσον η εγχώρια βιομηχανία δεν ορίζεται επακριβώ στο κείμενο της συμφωνίας, θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι σε περίπτωση που υπάρχει ζημία ή απειλή για ζημία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε μια, οι περισσότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βιομηχανία τους, και αυτό ενισχύεται και από πρόσφατα παραδείγματα. Έχουμε δει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει τέτοιε περιφερειακέ ρήτρε. Για παράδειγμα, στον ε, εφαρμοστικό μηχανισμό για τι περιφερειακέ συμφωνίε. Ακόμη και αν αυτέ καθεαυτέ δεν προβλέπουν περιφερειακή ρήτρα. Κάτι δηλαδή που προσωμιάζει με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την ε, Κορέα. Τώρα πέραν αυτών πρέπει να τονίσω και άλλα δύο σημεία. Πρώτον, ότι η ερμηνεία αυτή υπόκειται στι διευθετήσει επίλυση διαφορών τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Δηλαδή, η Κορέα θα μπορούσε να αμφισβητήσει τα όσα λέμε. Λέγοντα ότι εφαρμόζοντα περιφερειακή ρήτρα, κάνετε την ρήτρα αυτή πιο ευνοϊκή για εσά. Μπορείτε να την χρησιμοποιείτε πιο συχνά από ό,τι θα οφείλατε. Και έπειτα, δεν μπορεί κανεί να γνωρίσει το γεγονό ότι μια τέτοια περιφερειακή ρήτρα στην πράξη θα απορρίθμιζε την ε, εύρυθμη λειτουργία τη ενιαία αγορά. Για αυτού λοιπόν του λόγους, κατά τη δική μα νομική άποψη, αυτό που συστήνουμε είναι η Επιτροπή να προχωρήσει παρόλα αυτά με την περιφερειακή ρήτρα, εξασφαλίζοντας όμως ότι θα χρησιμοποιείται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και προσωρινά. Και ότι ισχύει κατά τρόπο που δεν θα απορριθμίζει την ε, ομαλή λειτουργία της αγοράς. Η βασική μας λοιπόν σύσταση είναι ότι μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ρήτρα, αλλά κατ' εξαίρεση. Θα πρέπει λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο να δούμε το θέμα της περιφερειακής ρήτρα. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Ελπίζω ότι τα εξήγησα επαρκώς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την νομική υπηρεσία για αυτήν την ε, τοποθέτηση που εξετάζει το θέμα της νομιμότητας της περιφερειακής ρήτρα. Υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής για τόσο μας επινομική υπηρεσία. Uh, Εάν όχι... Ναι, Πρόεδρε. Ίσως η νομική υπηρεσία θα μπορούσε να μας εξηγήσει τι γίνεται με τις περιφερειακές περιοχές και πώς αυτές χρησιμοποιούν αυτή τη ρήτρα. Υπάρχει δηλαδή κάποια ειδική διάταξη τελωνιακή ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς επειδή πλήττεται μια περιφέρεια ή μια χώρα θεσπίζει ειδικέ διατάξεις για, το, για τα τελωνία. Αυτό Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που έχουμε ότι πρέπει να ισχύει κατ' εξαίρεση. Διότι θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικά μέτρα για τα κράτη-μέλη ή για περισσότερα από εν, του ενός κράτη-μέλη λόγω ακριβώς της πρακτικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Διότι στο παρελθόν δεν έχει πραγματικά εφαρμοστεί. Πρέπει να ισχύσουν εξαιρετικοί λόγοι Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν το λόγο λέμε ότι πρέπει κατ' και προσωρινά να ισχύσει. Ευχαριστούμε. Άρα δεν αμφισβητεί την νομιμότητα. Ω προς τις πολιτικές αρετές της περιφερειακή Ρήτρα. Θα αποφασίσουν τα μέλη της Επιτροπής μας. Λοιπόν, νομίζω λογικό θα ήταν το λόγο να πάρει ο κύριος Φάβα, ο εισηγητή μας, ο κ. Ζάλμπα μάλλον, συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη εδώ της Επιτροπής μας με τους οποίους είχα πολλές και διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων μου... με βοήθησαν πάρα πολύ να ετοιμάσω την έκθεση αυτή. Πρέπει να διευκρινίσω ότι η έκθεση αυτή είναι μια επιτυχία όχι μόνο δικιά μου, αλλά όλων των συναδέρφων, όλων των πολιτικών ομάδων που βρίσκονται εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Επί της ουσίας. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες οι οποίες ε, βοηθάνε να διορθώσουμε κάποια τεχνικά λάθη που περιλάμβανε η έκθεση. Για παράδειγμα η 42 η οποία βοηθά όσον αφορά τροπολογία 4, την επιτροπολογία. Επίση, υιοθετήσαμε και την συμβαστική τροπολογία 6 για να ικανοποιήσουμε τι τροπολογίε ε, των ε, κ. Σαρνέθ και Σάιθ όσον αφορά τις έρευνες. Επίσης, δεχτήκαμε τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τον ορισμό των ε, άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων. Είναι οι τροπολογίες 44 της κυρίας Μουσκαντίνη, η 45 του κυρίου Σούστα, η 46 του κυρίου Μπένετ, και 47 του κ. Δεύρε. Πιστεύουμε ότι χρειαζόταν η διευκρίνηση αυτή για να μην υπάρχει πια κανένα περιθώριο παρεξηγήσεων. Όσον αφορά τώρα τη συμβαστική τροπολογία 5, είναι μια τροπολογία η οποία έχει να κάνει με αυτόν που ζητάει να ξεκινήσει μια έρευνα και αποφασίσαμε ότι να υιοθετήσουμε την πρόταση του κ. Φέλντερ που λέει ότι η βιομηχανία θα πρέπει να εκπροσωπεί το 25% τουλάχιστον για να ευθυγραμμιστούμε με τις ρυθμίσεις που υπάρχουν όσον αφορά το anti-dumping. Επίσης δεχτήκαμε και την πρόταση του κυρίου Λάγκεν να βάλουμε και μια εσωτερική advisory group ώστε να μπορεί και εκείνη να ζητάει την έναρξη έρευνας και έτσι να μπορούν και άλλοι φορείς που είναι βασικοί να ζητήσουν έρευνα. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες τώρα οι οποίες έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την αυτοκινητοβιομηχανία. Πρόκειται για την 79 και την 81. Μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας στον κανονισμό αυτό, στη ρύθμιση αυτή, να μην γίνεται διάκριση σε βάρος κανενός τομέα. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε και την αυτοκινητοβιομηχανία, τις εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις ε, απασχόλησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκουν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το θέμα λοιπόν των δασμών το εξετάζουμε από αυτή την οπτική γωνία. Στις ε, διατάξεις της συμφωνίας περιλαμβάνονται αρκετά θέματα που θέλαμε και εμείς να καλυφθούν για μη δασμολογικούς φραγμούς. Είναι 85 και 30 τροπολογίες που εμείς τις έχουμε βάλει σε αιτιολογική σκέψη. Γιατί πιστεύουμε ότι εκεί έπρεπε να βρίσκονται. Το ίδιο έχουμε κάνει και όσον αφορά την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Ο κύριος Σούστα και η κυρία Μουσκαρδίνη και ο κύριος Ρινάλντι ζήτησαν κάτι τέτοιο. Επίσης, έχουμε συμπεριλάβει στην αντιλογική σκέψη και την τροπολογία 43 του κυρίου Λάγκε, που πιστεύουμε ότι αποτελεί μια πάρα πολύ καλή λύση για το πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα τι τροπολογίε, οι οποίε τροποποιούν τι προθεσμίε, κατά τη γνώμη μου εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί τη διάρκεια των ε, μέτρων που προβλέπει η ρήτρα διασφάλισης έχουν ήδη συμφωνηθεί στη συμφωνία. Οπότε πρέπει να είμαστε συνεπείς και να καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τις τροποποιήσουμε. Οπότε η νομική υπηρεσία επέμεινε για το ότι αν τροποποιήσουμε τα άρθρα αυτά, είναι σαν να πηγαίνουμε κατά της συμφωνίας. Εμείς θέλουμε να σεβαστούμε την ε, νομική αυτή γνωμοδότηση. Τώρα υπάρχουν και άλλες προτάσεις που έχουν να κάνουν με τους παράγοντες όσον αφορά την ζημιά ή την υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχει ζημιά. Τα έχουμε συμπεριλάβει. Στη συμβαστική τροπολογία 7 φαίνεται ότι ο κατάλογο των παραγόντων που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εξαντλητικό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Επίση, έχουμε συμπεριλάβει και περισσότερες λεπτομέρειες για διάφορα προϊόντα τα οποία κατά την κατασκευή τους ένα μεγάλο μέρος τους κατασκευάζεται σε τρίτη χώρα. Είναι, υπάρχει ένα ποσοστό 5% που πρότειναν πολλοί και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα περιοριστικό. Όσον αφορά τώρα την πρόταση δημιουργίας μιας πλαταφόρμας online, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και έχουμε ακούσει τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τελικά καταλήξαμε στην πρόταση της του κύριου Λάγκε με τη συμβαστική τροπολογία 10 που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη όταν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα να δημιουργηθεί μια τέτοια πλατφόρμα κάθε φορά που τεχνικά αυτό είναι εφικτό. Θέλω τώρα να σας εξηγήσω τις απόψεις μου για δύο θέματα. Το ένα είναι για την, ε, τα μέτρα διασφάλισης σε περιφερειακό επίπεδο και το δεύτερο είναι η επιτροπολογία. Έχουμε ακούσει τα επιχειρήματα τη νομική υπηρεσία τώρα, οπότε θα σα μεταφέρω τι δικέ μου σκέψει για τι τροπολογίε που έχουν να κάνουν με τα μέτρα διασφάλιση σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι οι 59, 60, 61 και 62, όπω επίση και εκείνες που έχουν να κάνουν με το άρθρο 2 παράγραφος 1. Εδώ πέρα μιλάμε για το regional industry, για αυτή την έννοια. Ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε συζητήσει για την τελική αυτή ρήτρα. Όπως ακούσαμε την νομική υπηρεσία, όλοι, και λέει ότι αυτή η έννοια πηγαίνει κατά των όρων έκτακτων περιστάσεων. Οπότε εμείς προτείνουμε να επιμείνουμε στην αρχική μας τροπολογία 7 που αναφέρεται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Διασφάλισης και που ορίζει το περιφερειακό επίπεδο, ότι αποτελείται από ή από πολλά κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα την επιτροπολογία. Ο στόχο μα με την τροπολογία που προτείνουμε είναι ο εξή. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, ώστε να βρίσκεται επίση όρις με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε με τι διαπραγματεύσει μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Γι' αυτό, συνάδελφοι, πρέπει να εμείνουμε σε μια ισχυρή θέση εφόσον θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί τώρα έτσι έχουμε μια πιο γενική άποψη και δουλέψαμε από κοινού πολύ επικοδομητικά και θεωρώ ότι έχουμε συμφωνήσει σε 7 βασικά σημεία τα οποία υποθέτω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε αύριο. Πρώτο σημείο, θέλουμε οι κανόνες ε, να συμπεριλαμβάνονται και στο, στην ρήτρα διασφάλισης. Έχουμε μια ε, προσθήκη στο 3 με την ε, τροπολογία 29 και έτσι νομίζω ότι καθίσταται σαφές ότι θέλουμε αυτό να ισχύει πριν από την ε, θέση σε ισχύ. Ε, ειδικά στην ε, ρήτρα διασφάλισης. Δεύτερον, δεν θέλουμε να υπάρχουν δασμολογικά προσκόμματα στο εμπόριο. Τρίτον, θέλουμε και κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά στην συμφωνία τα οποία όμως θα πρέπει να μην ε, μετατραπούν σε ε, προσκόμματα προς τον ανταγωνισμό, επίσης σε ειδικέ οικονομικές ε, ζώνες. Όταν δηλαδή κάτι πρέπει να εφαρμοστεί με βάση συγκεκριμένα προϊόντα, θα πρέπει να ανανεώνεται η συμφωνία. Επίσης αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία, συγκεκριμένοι δείκτες, ενιαίοι δείκτες, άρθρο 5, ε, διαφάνεια μέσω της online πλατφόρμας. Έκτον, θέλουμε η κοινωνία των πολιτών η οποία έχει, έχει ε, λάβει μεγαλύτερη αξία μέσω αυτής της συμφανίας, μέσω των συμβουλευτικών ομάδων, να συμπεριληφθεί εδώ. Και έβδομον, φυσικά, θέλουμε η επιτροπολογία να είναι καθορισμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να παίξει πιο σημαντικό ρόλο. Αλλαγή λοιπόν της ε, διαδικασίας επιτροπολογίας, και αυτό που ζήτησε ο συνάδελφος Αρίφ και να αφήνουμε την τελευταία λέξη στο κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί αυτό θα αποτελέσει ίσως ε, και το πρότυπο για, τις, ε, για τη μελλοντική νομοθεσία. Οπότε χαίρομαι που καταλήξαμε τελικά στη συμφωνία για αυτά τα σημεία. Ένα σημείο έχει μείνει έτσι εκρεμές, το θέμα των περιφερειακών ρητρών. Ε, ακούσαμε ότι αν θα υπάρξουν καταρχήν θα υπάρξει μόνο αυτή η εξαίρεση που ανέφερε ο συνάδελφος στην, ε, στην τροπολογία 7 και που είναι του εισηγητή. Ίσως λοιπόν αυτό θα μπορούσαμε ακόμη να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω, αλλά γενικώ θεωρώ ότι επιτύχαμε να βάλουμε το Κοινοβούλιο στη θέση που του αξίζει. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστούμε, ο κύριος Καζάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ο κύριος Ζάλμπα, ο εισηγητής σας, και πολύ στενά με όλες τις πολιτικέ ε, πολιτικές ομάδες για την έκθεση Η θέση του, πιστεύω, εκφράστηκε σωστά με τις συμβαστικές μας τροπολογίες συνολικά. Συμφωνούμε περίπου σε όλα τα σημεία των συμβιβαστικών τροπολογιών. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τι προθεσμίε, συμφωνώ με την πρόταση ότι η διαδικασία έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί το περισσότερο σε μια προθεσμία για 200 ημερών αντί για 6 μήνε. Πρέπει να είναι μια ταχεία διαδικασία αυτή, γιατί πρόκειται για μια και μόνη χώρα. Και όσο για την περιφερειακή ρήτρα διασφάλιση, συμφωνώ με τον εισηγητή. Πιστεύω ότι η ιδέα να δώσουμε το δικαίωμα δράσης σε πολλά κράτη-μέλη που μπορεί να δράσουν ω περιφέρεια η περιοχή, είναι καινοτόμη, καινοτόμα, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, τοποθέτηση της νομικής υπηρεσία που μόλις ακούσαμε. Οπότε θα πρέπει τέτοια ρήτρα αν ισχύσει να ισχύει κατ' εξαίρεση και προσωρινά. Επίσης, για να υπάρχει σωστή ανταλλαγή ε, ε, πληροφοριών μεταξύ βιομηχανία και κοινοβουλίου. Θα συμφωνήσω επίση με την πρόταση του εισηγητή σχετικά. Και για τι διευκρινήσει του κυρίου Ζάλμπα για το είδο των οικονομικών φορέων νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη η τοποθέτησή του και κάνει τον κανονισμό πολύ πιο σαφή. Και για τα μέτρα επίβλεψης είναι σημείο κλειδί αυτό για την ομαλή διεξαγωγή των ε, εξαγωγών και εισαγωγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιας Κορέας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιοι είναι οι ευαίσθητοι τομείς που ενδεχομένως να πληγούν. Και το θέμα των δασμών για αυτή τη Συμφωνία Ελεύθερων Συλλαγών μας απασχολεί ιδιαίτερος αλλά είναι κάτι που ούτως ή άλλως διαρκώς το έχουμε μεταξύ των προτεραιοτήτων μας. Εδώ απαιτείται η εφαρμογή του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου για του κανόνε προέλευση, το θεωρώ απαραίτητο αυτό, και όσο για του κανόνε τη επιτροπολογία, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ακόμη και μετά την αναθεώρηση των διαφόρων εργαλείων μα, η εμπορική πολιτική θα παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ένωση. Επ' αυτού θα ήθελα μάλιστα να ακούσω και την άποψη του κυρίου Ζάλμπα, του εισηγητή και τη νομική υπηρεσία. Να μα πούν ποια είναι η τελική του τοποθέτηση για το σημείο αυτό. Αυτά είχα να πω. Βεβαίω, κάποιε τροπολογίε από τον ε, σκιώδη συγκεκριτή μα, τον κύριο Τόιρα και τον κύριο Ρινάλντι, έχουμε να τι εξετάσουμε ακόμα. Ελπίζω όμω ότι θα εγκριθούν, θα, τις, ε, θα συμφωνήσει και ο εισηγητή και θα εγκριθούν και από την Επιτροπή. Πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή, Εδώ έχουμε τον κύριο Στέρντι. Ναι, ήρθε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω δύο πράγματα να καλύψω. Πρώτα απ' όλα, κύριε Λάγκε, συμφωνώ για αυτό που λέτε όσον αφορά τις επιστροφές δασμών, το duty drawback. Όντως θα καταλήξουμε στο 1,5%. Οπότε, γιατί να μην δεχτούμε ότι μπορούμε να έχουμε τέτοιες επιστροφές δασμών. Πάντα με απασχολούσε, κύριε Ζάμπλο, το θέμα της ε, καταγωγής. Οπότε η ιδέα σας μου αρέσει. Ίσως θα μπορούσαμε να τη διευρύνουμε περισσότερο. Να μας πείτε πώς ακριβώς μπορείτε εδώ να συμπεριλάβετε διάφορες χώρες. Η έκθεσή σας πάντως είναι εξαίρετη. Συγχαρητήρια μπορούμε πραγματικά και κυριολεκτικά με όλα να συμφωνήσουμε. Το θέμα των περιφερειών, για παράδειγμα, είναι κάτι που το ζητούσαμε. Ωραία, λοιπόν, μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει, λέει ο Πρόεδρος, και θα ψηφίσουμε αύριο. Έτσι, κύριε Σιγητά, θέλετε τίποτα να προσθέσετε, μήπως. Απλώς και μόνο για τα μέτρα διασφάλισης σε περιφερειακό επίπεδο. Ορισμένοι, ορισμένες χώρες, ορισμένες ε, περιοχές, οι κλάδοι έχουν κάποιες ανησυχίες. Εγώ όμως θέλω να πω ότι θα κάνουμε παραπάνω προσπάθεια για να πείσουμε όσους έχουν κάποιες αμφιβολίες για τα κέρδη από αυτή τη συμφωνία. Τα ωφέλη. Και αυτό προσπαθούμε να το πετύχουμε και με τη μέτρα διασφάλισης σε περιφερειακό επίπεδο για την οποία θεωρούμε ότι είναι για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος. Ποιος ε, θέλει να προσθέσει κάτι για την Πετροπολογία, μου είπε η νομική υπηρεσία. Έχει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ. Αν θέλετε, να το κοιτάξουμε. Αν έχετε χρόνο, ευχαρίστως λέει η νομική υπηρεσία. Ουσιαστικά στηρίζουμε την προσέγγιση του εισηγητή με την τροπολογία που αναφέρεται σε συμβουλευτική διαδικασία αντί για διαχειριστική. Η μόνη δυσκολία μας είναι με την τροπολογία εκείνη η οποία αναφέρεται σε αρνησικυρία, σε βέτο από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποφάσεις προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ή να μην τεθεί σε εφαρμογή η ρήτρα διασφάλισης. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν με τον κανονισμό 91 για μέτρα που θα τίθεται σε ισχύ. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να εφαρμόζουμε την αρχή της επιτροπολογίας σε ρυθμίσεις όπως αυτή που εγκρίνουμε τώρα πρέπει να γίνεται μνήα των όσων αναφέρονται στην Συμφωνία Πετροπολογίας που δεν προβλέπει μέτρα άρνηση κυρίας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το κανονισμό 291 και προτείναμε να υπάρχει το droit de regard που σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εμποδίσει κάτι το οποίο αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω προ το παρόν πρέπει να ακολουθήσουμε την απόφαση τη Επιτροπολογία και ένα τέτοιο μέτρο δεν προβλέπεται προ το παρόν. Αυτό είναι το μόνο στοιχείο που μπορώ να σα δώσω από τη νομική άποψη. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι θέμα πολιτική απόφαση. Πρόεδρο, ωραία, θα το λάβουν υπόψη του διάφορε πολιτικέ ομάδε αύριο κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία. Στο σημείο 20 τώρα θα πάμε τη ημερήσιας διάταξη. Για την ουσία της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την Δημοκρατία της ε, Κορέας. Πολιτικά πρόκειται για μια διμερή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης για 10 χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, τον Ρόμπερ Στέρντι τώρα και από εκεί και πέρα επιτρέψτε μου Εγώ να επαναλάβω κάποια θέματα που ακούσαμε στα μέσα ενημέρωση τον τελευταίο καιρό, που τα μέσα ενημέρωση κατηγόρησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υπεύθυνο για το ότι πήγε για τον Νοέμβριο τον νωρίτερο η επικύρωση της συμφωνίας αυτής. Εμείς όμως δεν έχουμε καμία ευθύνη. Από την αρχή της διαδικασίας εμείς ξεκινήσαμε τις συζητήσεις με το Συμβούλιο. Οπότε, αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνο, αυτό δεν είναι το Κοινοβούλιο. Θα δώσω το λόγο λοιπόν τώρα στο Ρόμπερτ Στέρντι. Έμαθα ότι είναι για τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ρόμπερτ. Uh, Έχεις το λόγο. Πρόεδρε, όταν φτάνει κανείς στη δική μου την ηλικία δεν έχουν τόση σημασία τα γενέθλια. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Πάμπλο. Γιατί τα περισσότερα από όσα αφορούν τη δική μου την έκθεση έχουν συζητηθεί. Ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνατε για να γίνει πιο αποτελεσματική έκθεση. Είναι σημαντικό αυτό και συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι εδώ δεν είμαστε για να καθυστερούμε τα πράγματα. Θέλουμε να έχουμε μια σωστή γνωμοδότηση και να περάσει με το σωστό τρόπο ώστε να είναι ισχυρή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Νότια Κορέα. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι βιομηχανίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν τα απαραίτητα μέτρα, όπω είπε ο κ. Λάγκεν, για να εξασφαλίσουν ότι τα πράγματα βαίνουν καλώ. Ε, γιατί αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, Πρόεδρε, είναι ότι εδώ μιλάμε για μια σημαντική ε, γνωμοδότηση. Ξεπερνά τι ε, συμφωνίε ε, ελεύθερου εμπορίου, οπότε πρέπει να το κάνουμε, να κάνουμε το κάθε τι με το σωστό τρόπο. Η δική μου γνωμοδότηση είναι απλώς νομοδότηση ε, ε, συνένεσης, δεν τροποποιεί καθόλου το κείμενο, αλλά θα υποβάλω και ένα επεξηγματικό μνημόνιο, το οποίο θα σας αποσταλεί, θα αποσταλεί μάλλον σε όλους τους κοιόδης σήμερα. Και βεβαίως θα ακούσω τα σχόλιά τους για να τροποποιήσουμε το κείμενο ώστε να ε, συμπεριλάβουμε τις απαιτήσει ε, όλων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να εγκρίνουμε αυτή την ε, γνωμοδότηση και να πάμε στην επικύρωση όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Είναι καλή για την Κορέα, είναι καλή για την Ευρώπη, ωφελεί τους καταναλωτές, ωφελεί τις βιομηχανίες, αλλά η Ευρώπη και όλες οι βιομηχανίες στον κόσμο ε, αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Οπότε μια τέτοια έκθεση μπορεί να βοηθήσει. Βεβαίως εγώ περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας και σήμερα και στις επόμενες δύο εβδομάδες, ή τέλος πάντων όσο θα χρειαστούμε, για να μπορέσω να τροποποιήσω και το επεξηγηματικό μου σημείωμα. Αυτά, έτσι, Πρόεδρε, εν συντομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επειδή είναι η πρώτη έκθεση για αυτή την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, και υπάρχουν και άλλες που πρόκειται να εξεταστούν, συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει να είναι υποδειγματική η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Και υποδειγματική και η έκθεση. Ο κύριος Λάγκερ. Ευχαριστώ. Όντως, έχουμε μία ε, συμφωνία υπόδειγμα, οπότε θα πρέπει να την ε, δούμε πολύ προσεκτικά, ειδικά γιατί ε, είναι η πρώτη συμφωνία μετά την Λισαβόνα. Και βεβαίως έχει να κάνει και με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τη θέση του Κοινοβουλίου, η οποία ενισχύεται. Οπότε, φαντάζομαι ότι και σε μελλοντικές συμφωνίες θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε πιο ισχυρό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και να συμμετέχουμε πολύ περισσότερο και όχι μόνο στο τέλος να έχουμε έτσι μια, μια δυνατότητα να πούμε ναι ή όχι γιατί μπορεί να χρειαστεί να παρεκκλίνουμε. Αυτή η έκθεση έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα και θετικά σημεία, τα οποία ε, άπτονται και των εργαζομένων και των εργοδοτών και των βιομηχανιών, η πρόσβαση στην αγορά, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τη χημική βιομηχανία ή πρόσβαση στην αγορά σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Και κάτι άλλο που είναι επίσης πολύ θετικό είναι ότι σε αυτή τη συμφωνία είναι η πρώτη φορά που έχουμε κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία συμπεριλαμβάνονται ως υποχρεωτικά. Ε, ας πούμε πρότυπα ε, για την βιωσιμότητα, τις, ε, όπως υπάρχουν από τον ΟΗΕ. Τα χαιρετίζω και ελπίζω ότι και στο μέλλον να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα πρότυπα που υπάρχουν για την, από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Να δούμε τι γίνεται και με τα συνδικάτα. Κάποια παραδείγματα από το παρελθόν δείχνουν ότι αυτά τα βασικά δικαιώματα είχαν ε, τεθεί ένα αμφιβόλο. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό, αυτό το κίνδυνο μπορούμε να τον αποφύγουμε και αυτό είναι το θετικό στη συμφωνία. Και επίσης συμπεριλαμβάνεται και η κοινωνία των πολιτών και των ε, Κορεατών και η Ευρωπαϊκή. Γιατί έχουμε και αυτά τα εσωτερικά συμβουλευτικά όργανα με μη κυβερνητικέ οργανώσει, συνδικάτα και βιομηχανία. Οπότε όλοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τι γίνεται με αυτέ τι συμφωνίε τη Διεθνή Ελεύθερου Εμπορίου. Και αυτό είναι σημαντικό και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχίσει έτσι, γιατί έτσι μπορεί να συμπεριληφθεί και να συμμετέχει ω το δυνατόν περισσότερο και η κοινωνία των πολιτών. Τώρα, να σας πω πού βλέπω εγώ το ένα προβληματάκι. Ε, κατασκευές, ε, κλωστοφωτουργικά και αυτοκινητοβιομηχανία. Για τις κατασκευές, για, για την αυπήγηση, συγγνώμη, είχαμε προβλήματα στο παρελθόν με μέτρα για το, για το anti-dumping και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας έτσι ώστε, η βιομηχανία της ναυπήγησης εδώ να έχει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει μέλλον. αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό, ε, εδώ, ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί ο όγκος του ο εμπορικός, ε, όχι από τα αυτοκίνητα, αλλά λόγω αξίας είναι τεράστιος. Ίσως να είναι και μεγαλύτερος από άλλους τομείς. Και όντως εδώ θα πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα εάν Έχουμε ισότητα, ισοτιμία ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα εδώ που πρέπει να τεθούν. Ένα ερώτημα είναι γιατί οι Κορεάτες, οι κατασκευαστές, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ε, ανταλλακτικά ε, από τρίτες χώρε με τις οποίες δεν υπάρχει ελεύθερη, ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και δεν πληρώνουν φόρο, τελωνιακό φόρο, τελωνιακό δασμό. Και εμείς ή ξέρω εγώ μπαταρίες για τα... όταν αγοράζουμε μπαταρίες για τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρώνουμε τον τελωνιακό δασμό. Αυτά πρέπει να τα, να τα διασφαλίσουμε. Υπάρχει και η ρήτρα διασφάλισης για τα πέντε χρόνια. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συγκεκριμένε ρυθμίσει και σε αυτή τη ρήτρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό. Την ε, Παρασκευή μίλησα με έναν ε, ε, προμηθευτή από Ευρωπαίο, ο οποίος μου είπε ότι οι άλλες χώρες δεν, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τηρούν τις ίδιες προϋποθέσεις που τηρούν οι κατασκευαστές εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά σε ποιο, ε, σε ποιο βαθμό αυξάνονται αυτές οι εισαγωγές ή εξαγωγές των προϊόντων από τρίτες χώρες. Η αυτοκίνητο, αυτοκίνητο βιομηχανία στην Νότια Κορέα είναι πολύ μονοπωλιακή. Νομίζω ένα, μια εταιρεία έχει το 80% της αγοράς και φυσικά έχει και την απόλυτη δεσπόζουσα θέση. Ένα δεύτερο για την αυτοκίνητο βιομηχανία που δεν, δεν ε, αφορά την ε, επιδείνωση του ανταγωνισμού, αλλά έχει να κάνει με την πρόσβαση στην αγορά, στην Νότια Κορέα. Είναι πολύ μικρότερη βέβαια η αγορά, το ξέρουμε, δεν συζητείται αυτό, αλλά υπάρχουν εκεί πάρα πολύ σημαντικά προσκόμματα στην πρόσβαση. Ερώτημα λοιπόν. Τι γίνεται με τους μηχανισμούς πρόσβασης, τι γίνεται με τη φορολόγηση τι γίνεται με την νομοθεσία για το περιβάλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον και στα πλαίσια μιας συμφωνίας που θα έχει να κάνει με την πρόσβαση στην αγορά και θα την ανοίγει, να είναι σαφές, ότι δεν θα υπάρχουν δασμολογικά προσκόμματα, ε, στρεβλώσεις και ότι οι ευρωπαϊκοί ε, κανόνες θα αναγνωρίζονται, ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρυνση Ελπίζω να μπορέσει αυτό με κάποιο τρόπο να το καταστήσει πιο σαφέ στην έκθεσή σου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ε, ναι, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Συμφωνώ. Είναι η πρώτη συμφωνία για την ε, συμφωνία αυτή βάσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι και ω Ευρωβουλευτές και ω Επιτροπή για το διεθνέ Εμπόριο. Τροποποιώντας στέλνουμε κάποια σαφή μηνύματα που κατά τη γνώμη μου είναι δύο. Πρώτον, ότι είμαστε υπέρ των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, αλλά πρέπει να είναι ισορροπημένες και εφόσον είναι ισορροπημένες μπορούν να αποφελθούν από αυτές και δύο πλευρές. Έπειτα, όπως λέει και ο κύριος Λάγκε, πρέπει να στείλουμε ένα άλλο σαφές μήνυμα ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ακόμα περισσότερο. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. επόμενος, ο Μίτσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο πράγματα που είναι σημαντικά, παρόλο που συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο κύριο Λάνια. Ειδικά για τη σημασία αυτή τη πρώτη ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μετά τη Λισαβόνα. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Έχουμε την ε, οικονομική, τη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία έχει πλήξει πάρα πολλούς εργαζόμενους που εργάζονται ακριβώς σε αυτούς τους τομείς τους οποίους αφορά η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Οπότε πρέπει να τονίσουμε την αναγκαιότητα της τα οικολογικά κριτήρια, τα κοινωνικά κριτήρια για τις μελλοντικέ συμφωνίες και τη συνεργασία μας με την Κορέα στον τομέα του εμπορίου να, τους, να τα διασφαλίσουμε, να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Οπότε πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσουμε προσεκτικά, να δούμε πώς μπορούν να τηρηθούν οι κανόνες, έχουμε τις οδηγίες πλαίσιο για τα πρότυπα και πώς εφαρμόζονται. Γιατί αυτή η συμφωνία θα πρέπει να αναγνωρίζεται και από τους εργαζόμενους, γιατί αλλιώς θα συμφωνήσουμε εμείς σε μια στρατηγική, η οποία όμως θα ενισχύσει τις ε, ανισότητες μεταξύ των ε, εργαζομένων στην Ευρώπη και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να γίνει. Οπότε πρέπει να την πάρουμε πολύ σοβαρά αυτή την Συμφωνία Ελεύθερου Μπορείου και να την παρακολουθούμε πολύ στενά. Δεύτερον, πολύ σωστό, το είπε και ο συνάδελφος Στέρντι, ότι αυτή η συμφωνία είναι μια ε, συμφωνία εταιρική σχέσης. Οπότε διαπραγματευόμαστε επίσης όρις με τους Κορεάτες. Οπότε και το ενδιαφέρον της, ε, του, του, των πολιτών της Νότιας Κορέας πρέπει να ληφθεί υπόψη και βεβαίως και το ενδιαφέρον της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης. Η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε τέτοιες συμφωνίες, το είπε και ο συνάδελφος, είναι σημαντικό και πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στο να υπάρξουν τέτοια κοινωνικά πρότυπα σε χώρε με τι οποίε συνάπτουμε συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου, ώστε να μην υπάρχει dumping μετά στον ανταγωνισμό, αλλά με τους εταίρου μας από κοινού να μπορέσουμε να κανονίσουμε, να ρυθμίσουμε μία νέα οικονομική πολιτική. Αυτό συζητήθηκε και στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, για τη μελλοντική δηλαδή οικονομική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Εντάξει, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, παρόλο που υπήρξαν διάφορε αντικρουόμενε απόψει. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε πολύ προσεκτικά στη συζήτηση και γνωρίζοντα όλε αυτέ τι παραμέτρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά τη ρήτρα διασφάλισης. Δεν θα επιμείνω λοιπόν σε αυτό. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σάμπα και επίσης να συγχαρώ και τον κύριο Στέρντι για το έργο που μόλις ξεκίνησε τώρα. Για την περιφερειακή ρήτρα διασφάλισης, να πω τα εξή. Πρώτον, δεν συζητούμε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ή εταιρική σχέση ή διασύνδεση με μια φτωχή χώρα. Εδώ προσπαθούμε να καθορίσουμε μια συμφωνία με μια χώρα που έχει επιτύχει πρότυπα ποιότητας για, για το βιωτικό επίπεδο και για την ανάπτυξη που προσωμιάζουν πολύ με τα δικά μας. Εμείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε θύλακες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας και προβλημάτων πολύ μεγαλύτερους από ό,τι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Έπειτα, όταν προχωρούμε σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών πρέπει κάποιες φορές να περιμένουμε και 10 χρόνια. Κάποιες φορές εγώ έχω δει να περιμένουμε και 11 και 12 χρόνια. Εδώ μιλάμε για ένα ε, πλαίσιο πολυμερές σχέσεων, πολυμερών σχέσεων, το οποίο περνάει κρίση. Οπότε δεν μπορούμε να παρεμποδίζουμε τη σύναψη σχέσεων με μια συγκεκριμένη χώρα για να γίνει αυτό υπόδειγμα για τη σχέση μας με τους υπόλοιπους. Και όπως είπε ο συνάδελφος Λάγκε, όλες οι θετικές πτυχές θα πρέπει παρόλα αυτά να ακολουθούν κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Οι αρνητικές πτυχές από την άλλη θα έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις και για τον πληθυσμό το δικό μας και το βιωτικό τους επίπεδο. Τώρα, για την Κορέα και όχι για τη Ρουάντα, τι θα γίνει με, τις, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα εργασιακά τους πρότυπα, εάν εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θεωρήσουμε δεδομένο ότι συζητούμε με μια χώρα ισότιμη και περάσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς να διακριτήσουμε ότι είναι προφανές. Αυτά τα πράγματα για μια χώρα όπως η Κορέα είναι δεδομένα. Δεν θα ήταν δεδομένα ίσως για μια χώρα όπως η Κίνα ή η Ινδία. Όμως για χώρες όπως η Βραζιλία ή η Κορέα θα πρέπει να αρχίσουν να θεωρούνται δεδομένα. Τώρα, το μέρος που ίσως είναι αρνητικό ε, είναι τελείως δικό μας. Διότι αν εμείς αφαιρέσουμε από αυτή τη συμφωνία τις ε, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, διότι όταν μιλάμε για υπηρεσίες προσθέτουμε λόγια τα οποία προσπαθούν να εξηγήσουν στο κοινό το τι εννοούμε. Εδώ μιλούμε για το εμπόριο μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών. Ποινικοποιούμε ωστόσο το άνοιγμα των αγορών για την αγορά την κατασκευαστική. Διότι αν δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά του, δεν θα καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε τον οικονομικό αντίκτυπο τη αυτοκινητοβιομηχανία και τη κλωστοφαντουργία με τα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα που θα έχει το άνοιγμα των αγορών σε σχέση με την πώληση φαρμακών φαρμάκων ή κάποιου αλκοολούχου προϊόντο. Διότι περί αυτού ομιλούμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να πουλάμε στην Κορέα τυριά και λάδια δεδομένου του τι τρώνε και ποιε είναι οι διατροφικέ του συνήθειε. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να μιλάμε τη γλώσσα που καταλαβαίνει ο κόσμο. Ιδάλω, κάποια μέρα θα βρεθούμε στι εφημερίδε τι Ευρωπαϊκή στον τύπο, διότι καθορίζουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο το πώς θα πουληθούν οι μπανάνες, τα κολοκύθια και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τη στάση της Ευρώπης. Εδώ ε, ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, παρεμποδίσει τη συμφωνία με την Κορέα, γιατί θέλουν ακριβώς τη δική τους κατασκευαστική βιομηχανία να την εξασφαλίσουν. Αλλά δεν μιλάμε για την Κίνα και την Βραζιλία. Εδώ λοιπόν υπά... θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τον προστατευτισμό. Είμαι φιλελεύθερος σίγουρα σίγουρα στην οικονομική μου θεωρία. Όμω, δεν μπορούμε να μην είμαστε φιλελεύθεροι όταν από την άλλη έχουμε κάποιον φιλελεύθερο. Εγώ ως σοσιαλιστή νομίζω ότι πρέπει να έχω το μου και τους αρχέ τη κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη. Αλλά, άρα τα, τις κοινέ μας προδιαγραφές θα πρέπει να τις μοιραζόμαστε με άλλους, όχι με χώρες που τις θεωρούν δεδομένες και ούτε να ασκούμε την καταπίεση της πλούσιας δύσης στους φτωχούς όπως με τις χώρες ΑΚΕ. Όταν μιλάμε για την Κορέα και θέλουμε να εξασφαλίσουμε το χρηματοοικονομικό μας σύστημα και κάποιε ισχυρές βιομηχανίε, ας προσέξουμε γιατί υπάρχουν βιομηχανίε που δίνουν θέσεις εργασία, καλύπτουν τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά, την προστασία ε, για τον πληθυσμό της Ευρώπης. Σε αυτή την περίπτωση ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί δεν είναι δυνατόν μετά από μια δεκαετία να μην θέλουμε να συνάψουμε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με κάποιον. Αυτά, Πρόεδρε, ε, για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Κατά τα άλλα, μπορούμε σίγουρα να εργαζόμαστε για να αποσπάσουμε τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε για μια συμφωνία όπω αυτή. Όμω, α δούμε τι έκαναν και οι δημοκρατικοί τη Αμερική, των Ηνωμένων Πολιτειών για τα θέματα αυτά που έμειναν πάρα πολύ. Αλλά α μην περιμένουμε άδικα για μια συμφωνία η οποία θα έχει μόνο ακαδημαϊκή ισχύ και θα έχουν χαθεί μεταξύ εκατομμύρια θέσει εργασία στην Ευρώπη από τη δική μα την αναμονή. Ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα την Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι με το λίγο χρόνο που έχουμε χρειάζεται εδώ να μακρηγορήσω. Έτσι κι αλλιώ μα δόθηκε ευκαιρία πολλέ φορέ μέχρι σήμερα να συζητήσουμε για την συμφωνία αυτή και αύριο έχουμε και ακρόαση. Θα ξεκινήσω όμω με ευχαριστήσει προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη συμφωνία αυτή. Το γεγονό ότι συζητάμε και πριν ξεκινήσει η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης, νομίζω ότι αποδεικνύει την υπευθυνότητα με την οποία έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε η υπογραφή να γίνει το Σεπτέμβριο, να επικυρωθεί η συμφωνία αυτή το Σεπτέμβριο, οπότε να αποκορυφωθεί με τον τρόπο αυτό η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης. Τώρα πολλοί εδώ αναφέρθηκαν στη σημασία που έχουν οι μη δασμολογικοί φραγμοί. Οι συμφωνίες αυτές συνήθως έχουν ε, μεγάλα κομμάτια που αναφέρονται στην πειθαρχία όσον αφορά τους μη δασμολογικούς φραγμούς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά της Κορέας και γι' αυτό και θα γίνεται από κοντά έλεγχος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε η Κορέα να τηρεί τις υποχρεώσεις της. Σίγουρα θέλουμε να τηρούνται οι κοινωνικές προδιαγραφές και αυτό όχι μόνο εξαιτίας του εύρους της συμφωνίας, αλλά και επειδή τα συνδικάτα, οι βιομηχανίες και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις επίσης άμεσα θα συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων της Κορέας. Τώρα η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις. Φυσικά και θέλουμε να δούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει όσο γίνεται περισσότερο στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Εμείς θα είμαστε θετικοί και θα το δείτε και αργότερα στην ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε όσον αφορά την Ινδία. Θα το επαναλάβω αυτό και ευχαρίστω να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχουν οι ευρωβουλευτέ για τι εξελίξει των διαπραγματεύσεων αυτών. Πάντω, ακόμα θέλω να πω ότι δεν είναι ορθό να πούμε πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει μόνο μετά την ολοκλήρωση τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Δεν είναι αλήθεια αυτό διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει ψηφίσματα για τις διαπραγματεύσεις με την Νότια Κορέα και νωρίτερα με τον Ντέβιτ Μάρτιν, μάλιστα που ήταν εισηγητή για ένα τέτοιο ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό συμπεριλάμβανε συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα που θα έπρεπε να ληφθούν στις διαπραγματεύσεις. Με χαρά μπορώ να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό λάβαμε υπόψη μας τις συστάσεις αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν έλαβαν χώρα διαπραγματεύσεις αυτές. Από εκεί και πέρα Ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, με κάθε ευκαιρία ευχαρίστως να το συζητήσουμε και για ειδικού οικονομικούς κλάδους. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ανεξάρτητο ε, εμπειρογνώμονα να ελέγξει την ε, συμφωνία αυτή. Υπάρχει σχετική έκθεση και ό,τι ζητήματα μπορεί να θέσει η δικιά σας Επιτροπή κάποιος Ευρωβουλευτής εδώ για τη συμφωνία αυτή, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Πρόεδρο, ωραία. Κλείνει έτσι η ανταλλαγή απόψε. Το λόγο εισηγητή πάλι ο κύριο Στέρμπι. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λάγκε έθεσε κάτι που νομίζω ότι θα έπρεπε να διευκρινιστεί. Αναφέρθηκε στο αντι dumping Όσον αφορά εμένα, σε όλες τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕΜ, οποιαδήποτε χώρα και αν πρόκειται, υπάρχει νομοθεσία anti-dumping που μπορεί να ληφθεί υπόψη. Οπότε δεν χρειάζεται στην έκθεση, υπάρχει ήδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μου το επιβεβαιώσει ότι όντω έτσι είναι. Δεύτερον, όπως είπε και ο κύριο Σούστρα και άλλοι, θέλω να σα ακούσω. Κύριε Σούστρα, ξέρετε, πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για σας και εγώ είμαι υπέρ τη συμφωνία γενικά, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν πάντα να βελτιώνονται και είναι καλό για όλους μας να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Όλοι θα αποφεληθούμε, όπως και είπατε εσείς πολύ σωστά, κάποια θέματα ίσως χρειάζονται διευκρίνηση, αλλά η γνώμη μου είναι ότι η Ευρώπη μακροπρόθεσμα θα υποφεληθεί από μια τέτοια συμφωνία. Και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάμε. Το συνολικό όφελος για την Ευρώπη. Συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Και όντως σας ακούμε και θα συνεχίσουμε να σας ακούμε για ό,τι έχετε να πείτε στη, στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Βεβαίως και αυτό ισχύει για όλους φυσικά. Ευχαριστώ. Ε, μπορείτε, κύριε Γαρθία, να το διευκρινίσετε αυτό που ρώτησε ο συγητής, λέει ο Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, η συμφωνία με την Νότια Κορέα διασφαλίζει τα δικαιώματα και της Νότιας Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουν αντι-dumping. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός δεν υπάρχει συμφωνία, αλλά υπάρχουν διατάξει στη συμφωνία οι οποίες ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όσον αφορά το αντι-dumping. Πάντως η συμφωνία αυτή δεν περιορίζει με τίποτα το δικαίωμα ούτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε τη Κορέας να εφαρμόζουν διατάξεις αντι-dumping. Ακόμα και αν αποκλείεται από αυτή την διμερή συμφωνία. Πάντως ένας τομέας όπου η συμφωνία ξεπερνάει τους κανόνες της ΠΟΕ είναι επιδοτήσεις. Εδώ υπάρχει κάτι που ξεπερνάει τις διατάξεις του ΠΟΕ. Και μάλιστα είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τα ναυπηγεία, μια που αναφέρθηκε ο κύριος Λάγκη σε αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σας υπενθυμίζω ότι το σχέδιο έκθεσης θα το συζητήσουμε το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Μολδαβία. Η συγητής μας είναι ο Ιούλιος Βίνκλερ από το ΕΛΚΑ και πρόκειται για μια ανταλλαγή απόψεων πάνω στο σχέδιο έκθεσης του εισηγητή. Τον Ιούνιο, όπως ίσως ξέρετε, η Επιτροπή ενέκρινε μια απόφαση για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Μολδοβία. Για παρακολουθήστε εδώ λίγο, παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Και μην κάνετε φασαρία μέσα στην αίθουσα. Έλεγα λοιπόν ότι πρόκειται για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Μολδαβία ο, πρόκειται λοιπόν για κονδύλια μέχρι 19 εκατομμύρια ευρώ. Η αρρωγή αυτή είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπίσει η Μολδοβία την οικονομική κρίση. Αλλά επίσης και προκειμένου να ε, ενισχυθούν οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή. Ο συγκεκριτής μας έχει ήδη ετοιμάσει ένα σχέδιο έκθεσης το έχετε. Στα αγγλικά. Οπότε, ο Ιούλιος Βίνκλερ έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, uh, uh, είναι προφανές από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι συνάδελφοι ότι η Μολδαβία δεν είναι Κορέα. Αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, αναφέρω τρία πράγματα για την, ε, καταρχήν για την ε, συμφωνία που έχουμε, για τις τροπολογίες που προτείνω και για το χρονοδιάγραμμα. Πολύ σωστά είπατε, Πρόεδρε. Μιλούμε για τη μακροοικονομική χρηματική συνδρομή που είναι ένα δάνειο ουσιαστικά, 90 εκατομμυρίων ευρώ, σε τρεις δόσεις, φέτος, το 2010 και το 2011. Βοήθεια για μια χώρα που έχει περάσει πολύ δύσκολες ώρες τις τελευταίες δεκαετίες μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, μια χώρα που έχει δημοκρατική κυβέρνηση εδώ και 8-9 μήνες και η κυβέρνηση αυτή επιβεβαιώνει όποτε, σε όποια ευκαιρία και να της δοθεί την ε, ε, σύνδεση που έχει η χώρα αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, ε, για να δώσουμε τη συνδρομή πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια που να πληρώνται αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο πολύ σωστά επέλεξε να δείξει την στήριξή του στις προσπάθειες που κάνει η Δημοκρατία της Μολδαβίας. Βεβαίως, ε, συμφωνώ και με την πρόταση της Κομισιόν να δώσουμε στην ε, Μολδαβία αυτή την ε, συμφωνία. Ε, βεβαίως πρέπει να προτείνω κάποιες τροπολογίες γιατί πρόσφατα είχαμε μια τέτοια, ένα παράδειγμα τέτοιας συμφωνίας για μακροοικονομική χρηματική, χρηματική συνδρομή και το Κοινοβούλιο την συζήτησε κάποιε ανησυχίε που είχε σε ό,τι αφορά την ε, βελτίωση της διαφάνεια, τη αφήνεια και της λογοδοσία της ε, συνδρομής αυτή και επίσης το ρόλο του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της ε, βοήθειας. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω που είναι οι τροπολογίε. Πέντε τροπολογίες υπάρχουν. Η πρώτη και η πέμπτη αναφέρουν το θέμα της Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής ε, Επιτροπής ως εταίρου στην όλη διαδικασία και κατά την άποψή μου, ω συζητητού, η Κομισιόν θεωρώ ότι θα πρέπει τακτικά να μας ενημερώνει σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που αφορούν την ε, ε, συνδρομή και θα πρέπει να μας δίνει και τα απαραίτητα έγγραφα. Τροπολογία 2. Μια τροπολογία που αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει τακτικά να, χρηματο... να ε, πληροφορεί συγγνώμη, ε, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για τις εξελίξεις ε, στην, στην συμφωνία αυτή. Η τρίτη και η τέταρτη τροπολογία αφορούν το χρονοδιάγραμμα. Όπως και με την συμφωνία που είχαμε κάνει με την Ουκρανία, θέτουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την εκπλήρωση των όρων που απορρέουν από την συμφωνία αυτή για την συνδρομή. Αυτές είναι λοιπόν οι τροπολογίες μου. Και τρίτο σημείο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτό καθ' αυτό. 24 Ιουνίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες μεθαύριο. Ε, ε ψηφοφορία στην ΙΝΤΑ τον Ιούλιο, αλλά όχι τελική ψηφοφορία γιατί ακόμη θα πρέπει να γίνει η διαβούλευση και στα Εθνικά Κοινοβούλια ως ε, όρο που απορρέει από την Λισαβόνα και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και οι διαπραγματεύσεις με το, Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο και την Κομισιόν αν αυτές χρειαστούν. 30 ε, Αυγούστου είναι η συνάντηση της Επιτροπής μας και θα μπορούσαμε να κάνουμε την τελική ψηφοφορία αν όλα έχουν πάει καλά και 1η Σεπτέμβρη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την υποστήριξή σου, για την ε, δουλειά που έκανα και να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες και την γραμματεία πραγματικά για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν και με βοήθησαν στη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. <clears throat> και τώρα για το σχέδιο έκθεσης και τις τροπολογίες σας ξεκινήσουμε τη συζήτηση να δώσω το λόγο στον κύριο Κούτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει με την ε, δημοκρατία της Μολδαβίας στην Επιτροπή μας. Η αλλαγή στο πολίτευμα της δημοκρατίας της Μολδαβίας και το άνοιγμα Προ την Ευρωπαϊκή Ένωση τη χώρα αυτή θα πρέπει να είναι κάτι που θα το στηρίξουμε ω κίνηση. Ο υπουργό, ο κύριος Βλάντ Φιλάτ, δήλωσε πολύ ξεκάθαρα ότι ο σημαντικότερος στόχος της δημοκρατίας της μολδαβία για το μέλλον είναι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς. Οι διαπραγματεύσει ξεκίνησαν ήδη την 1η Ιανουαρίου 2010 Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι ότι η δημοκρατία της Μολδαβίας επλήγει ιδιαίτερως από την οικονομική κρίση και έχουν τεράστια δημοσιονομικά ζητήματα. Είναι μια χώρα με το χαμηλότερο κατά εισόδημα στην ε, περιοχή και εξίσου σημαντικό είναι ότι και ο συνασπισμός ο κυβερνητικός Ε, ο κυβερνητικό συνασπισμό δεν είναι αρκετά ισχυρό. Θα πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τη μακρονομική ενίσχυση για την ε, δημοκρατία τη Μολδαβία. Για να μπορέσουν και την οικονομία του να αναπτύξουν και να περάσουν σε δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει. Ο εισηγητή μα, ο κύριο ε, Βίνκλερ, είπε ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να συνεξεταστεί με τις προοπτικές της Ουκρανίας. Ως προς αυτό λοιπόν πρέπει να στηρίξω εδώ τον ε, εισηγητή μας στην τοποθετησή του. Είμαι υπέρ της γρήγορης έγκρισης αυτής της έκθεσης και της ε, έγκρισης του μακροοικονομικού αυτού μηχανισμού στήριξης της Μολδαβίας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σόλτς, μιας και βρίσκεται εδώ, έχει παρατηρήσεις. Ναι, Πρόεδρε. Σωστό είναι να έχουμε υπόψη μας την κατάσταση, την πολιτική που επικρατεί στην χώρα. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι φαινόταν. Εδώ και χρόνια, από όσο ξέρω τουλάχιστον εγώ, εδώ και έξι χρόνια, υπάρχει ένα σαφής ε, και της προηγούμενης κυβέρνησης προσανατολισμός σε πιο στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι με μια προοπτική για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν βέβαια επιθετική η πολιτική αυτή που είχε επιλέξει να ακολουθήσει η πρώην κυβέρνηση της Μολδαβίας. Σήμερα έχουμε το ε, αποτέλεσμα των πολλών εκλογικών διαδικασιών που έγινε. Τώρα έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση, έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ ασταθής. Οπότε ε, θα πω, ναι, εντάξει, η μακροοικονομική χρηματική συνδρομή άμεσα, αλλά όχι ως μέσο πολιτικής πίεσης, αλλά ως πραγματική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων που θέλουν να έχουν μια προοπτική στη χώρα αυτή, ε, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική ανάπτυξη στην Μολδαβία. Οπότε θα το ξαναμελετήσω εγώ το κείμενο, θα δω και τις τροπολογίες του εισηγητού και θα μπορούσα ίσως ε, να, έτσι, να προσθέσω και κάποια πράγματα στην έκθεσή του. Από την Κομισιόν, ο κύριος Τεμπράνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν θα ήθελε να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για την πρόταση, για τη συνεργασία μας, ε, για να επιταχύνουμε την διαδικασία έγκρισης. Η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί για να εφαρμόσει αυτή την πρόταση. Ελπίζουμε ότι με το παρόν χρονοδιάγραμμα θα καταφέρουμε να την εγκρίνουμε το Σεπτέμβρη. Για τις τροπολογίες τώρα, εμείς μπορούμε να ε, δεχτούμε τις τροπολογίες που θέλουν να συμμορφώσουν το κείμενο με όσα είχαμε ήδη συμφωνήσει με την Ουκρανία. Έχουμε παρεκκλίνει λίγο από το σχέδιο κειμένου γιατί η, η Επιτροπολογία συγγνώμη, αναφέρεται σε τέτοιου είδου ε, συμφωνίε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμεί προχωρούμε να δεχτούμε τι τροπολογίε που προτείνονται. Οι πιο πρόσφατε πληροφορίε που έχουμε για, τις, για, τη μακροοικονομική, για τις μακροοικονομικές εξελίξεις ε, είναι ότι μετά από αυτή την μεγάλη ύφεση ε, που έπληξε τη χώρα, το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προχωρά, ε, οπότε θεωρούμε ότι θα, θα ολοκληρωθεί η πρώτη αναθεώρηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, και θα δοθεί η επόμενη δόση των χρημάτων ε, τον Ιούλιο. Η κατάσταση πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητη όμως και σε ό,τι αφορά την φορολογική βιωσιμότητα γιατί πραγματικά η ύφεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και το πλήγμα που έχει δεχτεί η χώρα από την οικονομική κρίση είναι σημαντικό. Επίσης ε, η οικονομική κατάσταση είναι πολύ σημαντική. Η Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας έχει αναλάβει βεβαίω τα κατάλληλα μέτρα για να ε, σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση. Βεβαίως ε, περιμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα πέσει, προς το παρόν είναι αρκετά υψηλός. Οι προκλήσεις λοιπόν είναι πολύ σημαντικές και σε ό,τι αφορά τις διορθωτικές αλλαγές που δεν πρέπει να τις υποτιμούμε γιατί είναι σημαντικό να μπορέσουμε να, ώστε να είναι σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ε, μακροοικονομική συνδρομή το συντομότερο δυνατόν. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Okay, this our... Uh, Έτσι τελειώνει η συζήτησή μας για αυτό το θέμα. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 24 24η Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Και ερχόμαστε στο σημείο 7. Πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού 1215 του 2009 του Συμβουλίου. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο, συγγνώμη, έπρεπε να είχα δώσει το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Βίνκλερ, για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριος Βίνκλερ δεν ήθελα να σας διακόψω, όμω, έχω να πω δύο λόγια παρακαλώ, προκειμένου να κάνω μια παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ για τις νομοδοτήσεις που πήραμε. Σίγουρα ο κύριος Σελτίν καλείται από μας να υπογραμμίσει το ότι δεν θέλουμε να πιέσουμε, θέλουμε να στηρίξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι πρέπει να έχει γείτονες με σταθερότητα. Οπότε τέτοια θέματα όπως είναι η Μολδαβία ή η Ουκρανία είναι πολύ σημαντικά από αυτή την άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τις διαφορετικές αλλαγές εκεί για να στηρίξει τη δημοκρατία και όχι για να πιέσει. Ευχαρίστω να συζητήσω με όλους τους σκιώδους εισηγητές για να δούμε τι τροπολογίες θα μπορούσαμε να υποβάλουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρος. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα πάμε στο σημείο 7, τροποποίηση του κανονισμού αριθμός 1215 2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ε, εγώ ίδιος είμαι εισηγητής. Όπως ξέρετε, Στόχος είναι να επεκταθούν τα μέτρα του κανονισμού του Συμβουλίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου του 2015. Όπως θα δείτε και από το σχέδιο έκθεσής μου, εγώ δεν έχω αντιρρήσεις ουσιαστικά για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. συμφωνώ. Όμως, από τη στιγμή που ο κανονισμός περιλαμβάνει κάποιες εκτελεστικές εξουσίες που δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση επιτροπολογίας του 1999, γι' αυτό προτείνω κάποιες τροπολογίες ώστε να μπορέσουμε να ε, προσαρμόσουμε τους κανόνες στην κατεξοδότηση πράξης, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Προτείνω επίσης μια αλλαγή, να μην αποκλείεται το Κοινοβούλιο, αλλά να εφαρμόζεται η συνήθις νομοθετική διαδικασία για την έγκριση μέτρων προκειμένου να αλλάξουν, να διακόπουν ε, κάποια μέτρα βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού. Αυτές είναι οι κύριες πτυχές του σχεδίου μου έκθεσης που έχετε και στους φακέλους σας. Ξεκινάει η συζήτηση. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Ο Γιούλιος Βίνκλερ Να τα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θέλω να υπογραμμίσω ότι στηρίζει το ΕΛΚΑ την έκθεσή σας, το σχέδιο έκθεσή σας και τις τροπολογίες που προτείνετε. Κυρίως το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Με την τροπολογία αυτή και με άλλες ευθυγραμμιζόμαστε ουσιαστικά στη συνθήκη της Λισαβόνας και τίποτα άλλο. Πρόεδρος. Εκ μέρους της Επιτροπής, ο κύριος Φίλιπ Κουίσελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κόλεν Μπράουν ονομάζομαι και είμαι από την νομική μονάδα Διεθνούς Εμπορίου. Αντί για τον κύριο Κιούσο θα μιλήσω εγώ επειδή τα περισσότερα από τα σχόλια έχουν να κάνουν με την επιτροπολογία. Γι' αυτό μου ζητήθηκε εγώ να πάρω εδώ το λόγο. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας. Υπάρχουν δύο σημεία στα οποία θέλουμε να αναφερθούμε. Το ένα έχει να κάνει με την ουσία και το άλλο έχει να κάνει με τη διαδικασία. Όσον αφορά την ουσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με το περιεχόμενο ουσιαστικά των τροπολογιών, με το πνεύμα των τροπολογιών και συμφωνούμε, Επιτροπή εμείς, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στο νέο πλαίσιο που είναι εκείνο της συνθήκης της Λισαβόνας με τις διάφορες πράξεις όπου το Συμβούλιο ελέγχει η... τα κράτη-μέλη. Συμφωνούμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση όλων των πράξεων εκείνων που εγκρίνονται εκτός της διαδικασίας συναπόφασης. Όλες οι διαδικασίες επιτροπολογίας, ε, δηλαδή στον τομέα του εμπορίου. Τώρα όσον αφορά τις τροπολογίες, υπάρχουν ε, ορισμένα στοιχεία με τα οποία δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε. Για παράδειγμα, εμείς πιστεύουμε ότι για την τροπολογία 4 θα έπρεπε να είναι implementing act. Πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες 5 και 7 ήδη βασίζονται εκεί και υπάρχουν στις αποφάσεις για την επιτροπολογία. Επίσης έχουμε κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την τροπολογία 6 για το κατά πόσο πρόκειται για κατεξουσιοδότηση πράξη. Εμείς πιστεύουμε πως όχι. Επίσης σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 10 που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λάβει δράση, επίσης πρέπει να τροποποιηθεί. Οπότε, ναι, μεν συμφωνούμε με το πνεύμα, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες για συγκεκριμένες τροπολογίες που θα θέλαμε να συζητήσουμε ακόμα. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία. Στη δήλωση που επισυνάπτεται, είπατε κι εσείς Πρόεδρε ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η εμπορική προτίμηση για τα Δυτικά Βαλκάνια, για το Κωσυφοπαίδιο. Όπως γνωρίζετε, ο τρέχον κανονισμός εκπνέει στα τέλη της χρονιάς αυτής. Συνεπώς, πιέζει ο χρόνος και όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να φροντίσουν να έχουμε τον αναθεωρημένο κανονισμό που θα αντικαταστήσει τον κανονισμό αυτό. Επί της διαδικασίας λοιπόν προτείνουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Όπως ξέρετε και όπως αναφέρεται και στο επεξηγηματικό μνημόνιο στην πρόταση Επιτροπής, η Επιτροπή θέλει μια πρόταση όμνιμους που να τροποποιεί όχι μόνο αυτήν την πράξη αλλά και άλλες 23. Εμείς δουλεύουμε αδιάκοπα προκειμένου το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι. Και θα φροντίσουμε να ασχοληθούμε και με θέματα υπάρχοντα επιτροπολογίας. Θα φροντίσουμε και αυτό να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Η διαδικασία αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι έτσι τροποποιούνται όλοι οι κανονισμοί, μια και έξω, και προσαρμόζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας, με μια διαδικασία ad hoc. Επειδή πιέζει ο χρόνος, και πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να φροντίσουν να προχωρήσουμε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια καλύτερη προσέγγιση για να κάνουμε τις τροποποίησεις εκεί που χρειάζονται. Επί της ουσίας σας είπα ποιες είναι οι επιφυλάξεις μας. Πρόεδρος, ωραία. Ευχαριστούμε. Καταλαβαίνουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα λάβουμε υπόψη μας τη γενική αυτή πρόταση. Πάντως τώρα πρέπει να ξέρετε ότι δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε την έγκριση αυτής της ε, έκθεσης. Υπάρχει περιθώριο λοιπόν για συνεργασία μεταξύ μας, μεταξύ δηλαδή της Επιτροπής μας Διεθνούς Εμπορίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί και εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Οι τροπολογίες μου θέλουν να προλάβουν τα προβλήματα. Και ίσως προτίμασαν το έδαφος για να έχουμε την πρόταση αυτή για τη διαδικασία όμπνιμους από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Θα ανταλλάξουμε και πάλι απόψεις για αυτό το θέμα. Στι 10 Ιουλίου. Εννοούσα προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών, διορθώνει ο Πρόεδρος. Και περνάμε στο σημείο 8. Τροποποίηση του κανονισμού 1334 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίες διπλής χρήσης. Εισηγητής μας ο κύριος Λάιχτφριντ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το, αυτός ο φάκελος είναι πολύ σημαντικός και πολύ περίπλοκος και πολύ, με μεγάλες προκλήσεις. Έχουμε μία κατάσταση η οποία δεν μας ικανοποιεί. Και αυτό το κομμάτι που μπορούμε να αλλάξουμε με τη δική μας εργασία δεν είναι σε θέση να καταστήσει αυτή την ε, μη ικανοποιητική κατάσταση σε ικανοποιητική. Τι είναι αυτό που δεν μας ικανοποιεί. Υπάρχει το πρόβλημα του ότι τώρα ε, αυτά τα ε, προϊόντα διπλής χρήσης ε, στις εξαγωγές δεν ε, τη χάνουν της ίδιας μεταχείρισης από τις χώρες οι οποίες παράγουν τέτοιου είδους προϊόντα. Επίσης το όλο θέμα είναι λίγο αδιαφανές έτσι όπως το διαχειρίζονται και υπάρχουν και κάποια, κάποιες απώλειες στο σύστημα μεταξύ κομισιών και κρατών μελών κυρίως, αλλά και τώρα με το Κοινοβούλιο που θα πρέπει να εξηγενθούν. Προσπάθησα να εκπονήσω ένα έγγραφο εργασίας όπου ουσιαστικά χαρτογραφώ τα γεγονότα, ε, μπορεί κανείς να πει ότι θα πρέπει αυτή τη διαδικασία στο τέλος να την καταστήσουμε απόλυτα διαφανή. Θα πρέπει μέσω και της στρατηγικής της Λισαβόνας να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε όλο τον τομέα και θα πρέπει τώρα να δούμε ε, ποια επιτροπή είναι αυτή η οποία θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό και νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να είναι η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Και τέλος, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε, αυτές, σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι να μιλεί με μία φωνή. Ε, από όλη αυτή λοιπόν την ε, κατάσταση ε, είδαμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, ήρθαμε σε επαφή με, το, με τους σκιώδεις και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ίσως κόπιμο να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να προωθούμε τα πράγματα και σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν, αλλά σημαντικό είναι η Κομισιόν να υποβάλει μια τροποποιημένη πρόταση κανονισμού στο Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα στην Κομισιόν. Πόσο γρήγορα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμεί είμαστε τη άποψη ότι είναι απαραίτητο, απολύτω απαραίτητο να γίνει κάτι, να υπάρξει δηλαδή ένα νέο καθολικά νέος κανονισμός γιατί έχουμε τώρα αυτά τα α, παραρτήματα τα οποία ούτως ή άλλως τροποποιούνται και δεν μπορούν να μας λύσουν το πρόβλημα. Το ερώτημα τώρα είναι, είναι σκόπιμο το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να επεξεργάζεται την, κόμαση, την πρόταση Κομισιόν εάν μπορεί να σκεφτεί ότι η Κομισιόν θα υποβάλει νέα τροποποιημένη πρόταση. Και το Κοινοβούλιο υπό κάποιες συνθήκες θα μπορούσε να ψηφίσει, αυτή την, ε, νέα, θα μπορούσε να ψηφίσει με βάση αυτή τη νέα πρόταση της Κομισιόν. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα ήθελα να για τα οποία θα ήθελα να μου απαντήσει η Κομισιόν ώστε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, πόσο πρέπει να προχωρήσουμε τελικά. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να ξανασκεφτούμε τον κατάλογο των αγαθών ίσως και τον κατάλογο των χωρών, οι οποίες ε, πλήττονται από την απόφαση αυτή. Ε, προς τον παρόν είναι λίγο ανισόρροπη η κατάσταση και η πρόταση όπως έχει. Παρόλα αυτά, τίθεται το ουσιώδες ερώτημα. Καταρχήν, η Κομισιόν θα υποβάλει νέα πρόταση. Δεύτερον, θα υποβάλει γρήγορα νέα πρόταση, ώστε να μπορούμε να τη μελετήσουμε. Τρίτον, εμείς ως Κοινοβούλιο πώς μπορούμε να την υποχρεώσουμε με κάποιο τρόπο, να την αναγκάσουμε να το κάνει. Και όλα αυτά πώς μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Αυτά είναι τα ερωτήματα που έχω προς το παρόν και για τα οποία θα ήθελα μια απάντηση από την Κομισιόν. Τα ίδια ερωτήματα μοιράζονται και οι υπόλοιποι ε, ε, από τις ε, υπόλοιπε ομάδε. Οι υπόλοιποι συγκητές από τις ε, υπόλοιπες ομάδες. Θα ήθελα λοιπόν την απάντηση της ε, Κομισιόν. Όταν αποφάσισε η Επιτροπή μας να συνεισφέρει στη συζήτηση του θέματος αυτού με μια ε, γνωμοδότηση και έχουμε εδώ και τον κύριο Πατικόφερ ανέλαβε λοιπόν ο αρμόδιος συγκητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας αναφέρω πού έχουν φτάσει οι ως που έχουν φτάσει οι συζητήσεις στη Συναρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχω υποβάλει μια, ένα σχέδιο πρότασης. Οι συνάδελφοι των υπολείπων ομάδων έχουν υποβάλει τις τροπολογίες τους η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών έχει εκπνεύσει, οπότε σε αυτό τον τομέα θα μπορέσει να γίνει η συζήτηση. Στις συζητήσεις που έκανα εγώ με τους συζητητές, με τους κοιόδης συζητητές, διαπίστωσα ότι γενικώ μπορούμε να ακολουθήσουμε μια κοινή άγουσα η οποία έχει να κάνει κυρίως με την ασφάλεια. Δεν θα σας εκπλήξει αυτό που σας λέω και που θα βασίζεται στην αρχή ότι αυτά τα θέματα τα οποία όντως είναι πολύ ευαίσθητα δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στην ασφάλεια. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν συνολικά έχει κάνει έξι προτάσεις για τις εγκρίσεις γενικών εξαγωγών την οποία συζήτησε και η ομάδα στο Συμβούλιο στις 11 Ιουνίου και μεταξύ άλλων κατέληξε στο ότι μία από αυτές τις, ε, μία από αυτές τις έξι προτάσεις από αυτούς τους έξι τομείς ε, έχει να κάνει με τα κομπιούτερ και ε, τα αναλώσιμα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις αποστολές χαμηλής αξίας. Για αυτό το σημείο τα κράτη-μέλη στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου αναγνώρισαν ότι υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Οπότε, θα, σε σχέση με αυτό που είπε και ο συνάδελφος Λάιτφριντ, θα, θα ρωτήσω και εγώ το ίδιο την Κομισιόν. Μήπως θα μπορούσε η Κομισιόν σε σχέση και με αυτά τα νέα αποτελέσματα του Συμβουλίου να επεξεργαστεί αυτό που θα υποβάλει τελικά και παρά την εργασία του Συμβουλίου η Κομισιόν πιστεύει ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα και επίση το δεύτερο ερώτημα του συναδέλφου Λάιχτφριντ. Αν η Κομισιόν κάνει κάτι τέτοιο, πότε θα το κάνει. Άλλη μια παρατήρηση που, έχει να κάνει, που δεν έχει να κάνει μάλλον με τη ρύθμιση αυτή καθ' αυτή, αλλά έχει να κάνει με το πρακτικό της υπόθεσης. Είναι το πώς η κατάλληλη εφαρμογή μιας τέτοιας ρύθμισης μπορεί να εξασφαλιστεί. Γιατί απλώς εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι στις ΕΠΑ όπου το Υπουργείο ε, Εσωτερικών και Ασφάλειας είναι υπεύθυνο για τέτοια θέματα, ε, υπάρχουν χιλιάδες υπάλληλοι οι οποίοι ασχολούνται ακριβώς με αυτό, με τους ελέγχους εξαγωγών και κατά τη δική μου άποψη μέχρι τώρα δεν είναι απολύτως σαφές αυτό πώς θα γίνει με, τις, με τα κράτη-μέλη τα δικά μας και με τις δικές τους ε, τελωνιακές αρχές. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Η δική μου προσέγγιση και η δική μου εμπειρία με το θέμα ε, ακολουθεί και τις ε, σκέψεις που έρχονται από το Συμβούλιο. Ότι δηλαδή υπάρχει αρχή ε, που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για το επίπεδο ασφάλειας. Και από αυτό απορρέουν τρία βασικά ερωτήματα και τελειώνω πρόεδρε. Το ένα είναι αυτό που είπε και ο κύριος Λάιχτφριντ, το θέμα της, ε, του προορισμού αυτών των εξαγωγών, ο κατάλογος δηλαδή των χωρών που προτείνεται από την Κομισιόν είναι πραγματικά πολύ μακρύτερος από τον κατάλογο των χωρών που προτείνει το Συμβούλιο. Και εγώ θα ήμουνα υπέρ του να ακολουθήσουμε μια πιο προσεκτική άκουσα, αυτή δηλαδή του Συμβουλίου. Δεύτερον, είχα πει ήδη ότι υπάρχουν επιφυλάξεις σε σχέση και με τα low value shipments και τις σχετικές εγκρίσεις για τις ε, αποστολές χαμηλού κόστους. Εγώ είμαι της άποψης ότι μιλούμε για ποιότητα εδώ και όχι για ποσότητα και θα, ή θα έπρεπε να μιλούμε για ποιότητα και όχι για ποσότητα και σε ό,τι αφορά την ε, αξία. Αν ε, υποτιμήσουμε αυτές τις εξαγωγές θα, μπορούσαν, ε, θα μπορούσε να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ο οποίος μπορεί να δεν μετακυλείται κατά ανάγκη στην τελική τιμή του προϊόντος και ίσως κάποιες χώρες να αποτελέσουν και αντικείμενο επιθέσεων όπως έχει γίνει και το ΝΑΤΟ θα πρέπει αυτό να το πάρει υπόψη του. Και τρίτον, θα πρέπει να γίνεται και μία αναφορά εξάντε, εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους, ευχαριστώ και για τις πολύ καλές συζητήσεις που κάναμε. Το θέμα αυτό της διπλής χρήσης ε, είναι ένα όντως πολύ σημαντικό ζήτημα. Μιλούμε για προϊόντα τα οποία έχουν αξία για τη δική μας βιομηχανία, τα οποία όμως ε, χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο και καταλήγουν σε λάθος χέρια και μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες ζημιές. Θα ήθελα η Κομισιόν να μας εξηγούσε γιατί πιστεύει ότι το κείμενο που μας υποβάλλει είναι το σωστό εγώ είμαι τη άποψη ότι θα μπορούσε, ίσως, η Κομισιόν, όπως και ο συνάδελφος Λάκτφριντ το προτείνει, να μας υποβάλει ένα νέο κείμενο. Και δεύτερον, θα ήθελα επίσης πληροφορίε από την Κομισιόν για το ουσιώδες θέμα του τι θα γίνει με τους ε, υπαρχόντες κανονισμούς και πώς αυτοί θα εφαρμοστούν. Γιατί έχω την εντύπωση ότι οι υπάρχοντε κανονισμοί ε, εφαρμόζονται με τελείω διαφορετικό τρόπο από τα κράτη-μέλη. Γιατί λαμβάνω πολλέ ε, πληροφορίε από διάφορε επιχειρήσει διαφόρων χωρών που λένε ότι κάποια προϊόντα, όταν ας πούμε μιλούμε για μια, γερμα... μια εταιρεία με γερμανική έδρα, ε, λαμβάνουν πολλά, ε, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ε, να πάρουν εγκρίσει κτλ. Όταν αυτό το προϊόν θέλουν να το, κάνουν, να το εξάγουν με κάποια άλλη χώρα στο εξωτερικό, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να λάβουν αυτή την έγκριση. Οπότε είμαι της άποψης ότι αν ο κανονισμός προχωρήσει έτσι, θα πρέπει να τον δούμε γιατί η εφαρμογή και ο τρόπος εφαρμογής είναι πολύ διαφορετικός από κράτος σε κράτος και αυτό έχει μεγάλη, μεγάλες πολλές συνέπειες στα κράτη-μέλη και στις βιομηχανίες τους. Οπότε θα πρέπει ο κανονισμός αυτός να τον επεξεργαστεί η Κομισιόν και θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν τι θα γίνει τελικά με την εφαρμογή των κανονισμών στην πράξη, κατά πόσο μπορούν να εφαρμόζονται ενία σε, όλο το, σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα κρατημέλη και κατά πόσο υπάρχουν ε, κάποια σημεία κριτικής ε, που έχουν αποστείλει ίσως ε, οι βιομηχανίες στα κρατημέλη προς την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε λοιπόν την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου που ανέλαβαν το εγχείρημα να περάσουν σε ένα τόσο πολύπλοκο θέμα. Εδώ βρισκόμαστε στα όρια μεταξύ των ζητημάτων ασφάλειας και των εμπορικών στοιχείων. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο το εγχείρημα του εισηγητή. Θα συμφωνήσω πολύ μου σε σα για τα θέματα της ενιαίας αγοράς. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο, στην οριακή γραμμή μεταξύ ασφάλειας και των ε, μεριμνών των εμπορικών. Εδώ εμπλέκεται σαφώς η ενιαία αγορά. Τι θα γίνει λοιπόν με τον έλεγχο. η έλεγχη για τα θέματα ασφάλειας από το παρελθόν, από το 1995, βασίζονται στις αποφάσεις των 100 μελών, τι εξατομικευμένε. Το 10 αποφάσισε το 95 ότι εδώ μιλάμε για κοινή εμπορική πολιτική. Άρα η συνιστόσα της ασφάλειας στην απόφαση αδειοδότησης ενός προϊόντος δεν θέτει το ζήτημα αυτό, τη διαδικασία αυτή εκτός εμπορικής πολιτικής. Γι' αυτό επεξεργαστήκαμε τον κανονισμό που έχετε και τώρα μπροστά σας. Έχουμε μια διαδικασία εδώ οικοδόμηση της ενωσιακή διάσταση από του είδους τα θέματα. Για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου, συμφωνώ απολύτως, θέλαμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις και στο Κοινοβούλιο και ακούσαμε προσεκτικά όσα είπατε. Για το πρόβλημα που έχει να κάνει με την διαφορετική εφαρμογή των, των διαφόρων κρατών μελών ως προς τον ίδιο κανονισμό, οπότε πώς εξασφαλίζουμε έτσι την καλή ε, εφαρμογή. Υπάρχουν αρχές αδειοδότησης εδώ, οι οποίες αποφασίζουν αν θα εγκρίνουν κάποια προϊόντα ή όχι βεβαίως. Υπάρχει κατάλογος αντικειμένων ειδών τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας για όλους τους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά έχουν συμφωνηθεί σε διεθνέ επίπεδο και σε διάφορα καθεστώτα και κατηγορίε. Υπάρχουν όμω και άλλα προϊόντα για τα οποία τα κράτη-μέλη αποφασίζουν βάσει τη δική του διακριτική ευχέρεια εάν θα δώσουν εξαγωγικέ άδειε ή όχι. Υπάρχουν ανταλλαγέ απόψεων και συζητήσει σχετικά αλλά εδώ να απαντήσω και σε μια άμεση ερώτηση. Είχαμε παράπονα από εταιρείε που εξάγουν απευθεία σε τρίτε χώρε ότι είπαν ξέρω ότι δεν θα φτάσουν στον, τελικό χρήστη, στον ίδιο τελικό χρήστη τα ίδια προϊόντα, ενώ οι ανταγωνιστέ μου από ένα άλλο κράτο μέλο μπορούν να τα στείλουν σε αυτόν τον τελικό χρήστη, σε εκείνη τη χώρα. Έτσι λοιπόν δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία αλλά και με τη σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών. Έχουμε κάνει και κάποιε επισκέψει σε κάτι μελη για να δούμε ότι το σύστημα ισχύει παρομοίω παντού. Όμω δεν είναι απλή η προσπάθεια. Και ε, βεβαίω επαφιόμαστε και στην ε, ενίσχυση του Ευρωκοινοβουλίου εδώ. για το ζήτημα του κατά πόσον αυτή είναι η σωστή πρόταση και γιατί έχουμε αυτόν τον κατάλογο και όχι έναν άλλο, να πω ότι η πρόταση αυτή βασικά στηρίζεται στο τι έχουν τα κάτι μέλη ως εθνικές ε, αρχές ε, εξαγωγών, αδειοδότησης εξαγωγών. Υπάρχει δηλαδή ένας εμπειρογνώμων αδειοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχουν και διάφορες εθνικές, ε, εθνικοί φορείς στα διάφορα κράτη-μέλη. Οι εξαγωγεί λοιπόν από το κράτο μέλο Α μπορούν ελεύθερα ένα κατάλογο προϊόντων να τον εξάγουν προς ένα συγκεκριμένο προορισμό. Δεδομένου ότι υπάρχει βεβαίω ε, βάση σε αυτό το κράτος μέλος. εταιρείε δηλαδή στο κάτω μέλος Β. Έχουμε πάρει λοιπόν αυτές τις εθνικές αρχές, του εθνικούς φορείς και προσπαθούμε να τους συνενώσουμε σε ένα κοινό παρονομαστή. Αυτό είναι και η ουσία της πρότασής μας. Οι ανησυχίες ασφαλείας κάποιων κατωμελών μελών δεν είναι αναγκαστικά ανησυχίες που συμμερίζονται και άλλα κράτη-μέλη. Λόγω χάρη, οι, οι αποστολές ε, χαμηλής αξίας, low value shipments, σε δύο συγκεκριμένα κατημέλη, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αδειοδοτήσεις ε, χαμηλή αξίας σε εθνικό επίπεδο. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές οι εθνικές, ε, αυτοί οι εθνικοί χαρακτηρισμοί του Ηνωμένου Βασίλειου και της Γερμανίας μπορούν να ισχύσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ μιλάμε βέβαια για αξία περιορισμένη σε συγκεκριμένο αριθμό χωρών. και για φορείς που μόνο υπό τον τελωνιακό κώδικα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δικασία. Πρόεδρος, μπορείτε να συντομεύετε. Ναι, ένα τελευταίο σημείο για το εάν πρόκειται η Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση. Αυτή τη στιγμή μελετούμε το πώ θα διαμορφωθεί στο μέλλον η εμπορική μας πολιτική. Θα έρθει μια ανακοίνωση μετά το καλοκαίρι, όπως ξέρετε. Δεν μπορώ λοιπόν να προδικάσω τίποτα. Η πρόταση απλώς τη επιτροπή, θα ήταν η Επιτροπή σα να επεξεργαστεί την πρόταση αυτή, να προσπαθήσει να την εγκρίνει, γιατί σε κάθε περίπτωση είναι μια πρόταση που πηγαίνει στην κατεύθυνση που μα ε, διέγραψε και ο εισηγητή. Στην κατεύθυνση τη εσωτερική αγορά. Είναι λοιπόν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα παρακολουθήσουμε στενά τις συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να τραβήξει αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα να συζητήσω συγγνώμη από την Κομισιόν εάν δεν ήμουν σαφή την πρώτη φορά που πήρα το λόγο. Αλλά αυτό που αποκόμισα εγώ από τις ε, συζητήσεις με τους Κιώδης είναι μία, ότι υπάρχει, δεν υπάρχει θέληση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ε, επί αυτού του κανονισμού αν δεν υπάρχει προπτική για έναν γενικό κανονισμό. Και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που τίθεται και Δεν με ικανοποίησε απόλυτα η, η απάντησή σας και ο συνάδελφος Κάσπαρη επίσης συμφωνεί μαζί μου. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε λίγο αν μας λέγατε κάτι παραπάνω. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που είναι προς όφελος όλων. Και θα συμφωνήσω και με αυτά που είπε ο συνάδελφος ειδικά σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές. Γιατί ακόμη και αν υπάρχει ένα σύστημα οπλικό, όλα έχουν να κάνουν με κάποιο σύστημα πληροφορικής. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δούμε. Όπως είπα, αυτό είναι το σημαντικό που δεν έχει απαντηθεί από εσάς. Θα ήθελα να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ. Επιτροπή. Έχετε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Εάν η ερώτηση είναι εάν θα προτείνετε νέο κανονισμό το ερχόμενο δίμηνο ή τρίμηνο ή όχι, η απάντηση είναι όχι. Ακόμη βρισκόμαστε σε συζητήσεις. Πρόεδρε, πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, είμαι υπεύθυνο των σχέσεων με το Ευρωκοινοβούλιο. όλοι οι εκκρεμείς κανονισμοί έχουν υποβληθεί ξανά στην αρχική τους μορφή. Διότι συζητήσαμε με το Ευρωκοινοβούλιο και υπήρξε και έτοιμο από δική σας πλευράς να δείτε την αρχική μορφή στην αρχική τους μορφή της νομοθετικής προτάσεις, διότι έγινε κάποια δουλειά στο Συμβούλιο για πολλούς από τους κανονισμούς, όμως μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου πετύχαμε αυτή τη συμφωνία για τις κανονισμούς που αφορούσαν τη Γενική Διεύθυνση Trade. Να τους δείτε στην αρχική τους μορφή. Ωραία λοιπόν. Η εξέταση του σχεδίου έκθεσης της 30 Αυγούστου. Μετά την καλοκαιρινή διακοπή. Πάμε τώρα στο σημείο 9 νέα συζήτηση για την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Τη θεωρήσαμε δεδομένη, αναγκαία μάλλον αυτή, επειδή υπήρξαν αρκετέ δυσκολίε με αυτό το θέμα. Από το 2005 έχει επιτελεστεί ελάχιστη πρόοδο στο Συμβούλιο. Και πρόσφατα η επίσκεψη τη αντιπροσωπεία μα στην Ιταλία τον Μάιο συνέλεξε κάποιες ε, αντιδράσεις επιτόπου για το ότι είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί γρήγορα αυτό ο κανονισμό. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Μουσκαρντίνη, η οποία είναι αντιπρόεδρο τη Επιτροπή μα και κάθεται στα αριστερά μου, για να μα παρουσιάσει τι πρόσφατε εξελίξει. Κριστιανά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων νομίζω και ελπίζω ότι θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη και καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας για τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε. Το Ευρωκοινοβούλιο, όπως όλοι γνωρίζουμε, πριν από λίγους μήνες, κατά μεγάλη πλειοψηφία, τοποθετήθηκε θετικά στην έγκριση κανονισμού για την ένδειξη χώρας καταγωγής αυτό μετά την θέση σε ισχύ της Λισαβόνας έδωσε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Επίτροπο να αναθέσουν στην Επιτροπή μας να ξαναδούν στην όλη του εξέλιξη τον κανονισμό του 2005, τον περιβόητο αυτόν κανονισμό. Έτσι λοιπόν, τι περιμένει από εμάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εντοπίσουμε τα σημεία αυτά όπου ενδεχομένως ο κανονισμός θα πρέπει ελαφρώς να ανθρωποποιηθεί σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί στο μεταξύ. Ο κανονισμός είναι ένας κανονισμός που είναι ε, ιδιαίτερα επίκαιρος. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσει των πολιτών και των καταναλωτών των ε, ευρωπαϊκών κρατών και διασφαλίζει το δικαίωμά τους που από καιρό αναγνωρίζεται στους καταναλωτές και πολίτες ε, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Κίνας, του Καναδά και ούτω καθεξής. Θέλουμε να καθορίζει ο κανονισμός την ελευθερία επιλογής και την ελευθερία πληροφόρησης των καταναλωτών υπό την έννοια ότι περισσότερη ενημέρωση σημαίνει και περισσότερη δημοκρατία. Δεν θα ήταν σωστό να συνεχίσουμε να κρατάμε εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέση κατώτερη και υποβαθμισμένη σε σχέση με καταναλωτές της χώρας με σχέση με τους καταναλωτές χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και χωρών πιο καθυστερημένων όπως η Κίνα. Θέλουμε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ισότιμοι τουλάχιστον με τους Αμερικανούς. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθεί κάποια συμφωνία. Το Κοινοβούλιο λέει με τρόπο ξεκάθαρο στο Συμβούλιο ότι εδώ είναι αναγκαία να βρεθεί κάποια συμφωνία. Ιδάλω τα λόγια μα παραμένουν κενά ε, νοήματο. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών και την ελευθερία επιλογή. Ιδάλλω δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα. Θα λέμε μόνο λόγια στον αέρα. Αυτή είναι η δική μα λοιπόν θεώρηση των πραγμάτων. Τώρα, σε αυτό το σχέδιο έκθεση που σα έχω υποβάλει, θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε και κάποιες επιπλέον σκέψεις και θα ήθελα να επιμείνω στα εξή σημεία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές χώρες στον κόσμο, από το 1930 έχουν ανάλογο κανονισμό. Κανονισμό για όλα τα προϊόντα που μπαίνουν στο έδαφος τους στη χώρα. Ο κανονισμός που τώρα υποβάλλουμε και μας έχει υποβάλει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει μόνον ορισμένα προϊόντα. Διότι Θέλουμε να φτάσουμε στην έγκριση του κανονισμού χωρίς ε, διαγραφές και να τηρήσουμε τους χρόνους σεβασμού και συμμόρφωσης με τους κανόνες του κανονισμού, τις διατάξεις του κανονισμού, από όλες τις χώρες, χωρίς να έχουμε θέματα διαστρέβλωσης ή προβλήματα στα προϊόντα των εταιριών μας. Τώρα, από εμπορική άποψη, θεωρήθηκε πάντοτε ισότιμο και εύστοχο κάποιε σημαντικέ χώρε, όπω αυτέ που προανέφερα, να έχουν ένα σύστημα κανόνων για την ένδειξη χώρα καταγωγής ε, των προϊόντων που μπαίνουν στο έδαφο του. Για αυτόν τον λόγο η Ευρώπη, κάποιε ευρωπαϊκέ τουλάχιστον χώρε, δεν θα έπρεπε να έχουν πλέον αμφιβολίε. Αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε να τονίσουμε είναι ότι Η τροποποίηση που θα προτείνουμε και εμείς με τροπολογία αφορά το σημείο του κανονισμού που λέει ότι ε, στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νέες αναφορές, συμπεριλήψεις δηλαδή, προστίκες στον κατάλογο ή διαγραφές από τον κατάλογο του κανονισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι για τις νέες εμπορικές κατηγορίες, ε, για τη διαγραφή από τις ε, εμπορικές κατηγορίες που ήδη υπάρχουν, θα πρέπει να γίνονται μέσω του έργου της ανάλογης κοινοβουλευτικής επιτροπής. Διότι αυτό είναι έργο όχι μόνο τεχνικό αλλά πολιτικό κατά κύριο λόγο. Και την πολιτική συνιστόσα, ιδίω μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, την αναλαμβάνει όλο και περισσότερο το Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίω υπάρχει διάθεση συνεργασία και επικοινωνία με την Επιτροπή, κατά τρόπο ώστε να μην υπάρξουν ε, διαφωνίε, όμω ε, η αρμονική συνεργασία που ανέκαθεν υπήρχε θα πρέπει να συνεχιστεί και να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή να πείσουν το Συμβούλιο, όταν ενδεχομένω το Συμβούλιο δεν έχει αρκετό χρόνο να μελετήσει επαρκώ κάποια ζητήματα, οπότε δεν είναι και σε θέση να τοποθετηθεί ευνοϊκά. Επ' αυτού, και για να μην μακρηγορήσω, εφόσον έχω αποστείλει και ένα σχέδιο κειμένου για να καταλάβετε καλύτερα το θέμα, δεν θα μακρηγορήσω λοιπόν, Θα ήθελα απλώς να σας ζητήσω να συνεξετάσετε όλα τα θέματα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν και να έχετε υπόψη ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να τοποθετηθεί πλέον το Σεπτέμβριο. Ο χρόνος πιέζει και θα πρέπει κάπου να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στις υπόλοιπες γλώσσες πέραν των Ιταλικών. Ανοίγουμε λοιπόν την συζήτηση και δίνω το λόγο στον κύριο Σούστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Κριστιανά. Με συγχωρείτε Πρόεδρε να διακόψω και να πω ότι λυπάμαι, ξέχασα να πω προηγουμένως. Ε, ξέχασα να πω ότι το κείμενο έχει μεταφραστεί μόνο στα αγγλικά. Και αυτό με δική μας εσωτερική πρωτοβουλία. Να πω, θα ήθελα τα μέλη της Επιτροπής που νομίζω έχει προσλάβει κάποια άτομα τον τελευταίο καιρό. Θα έπρεπε να φροντίσει λοιπόν η Επιτροπή μας να καλύψει και τις μεταφράσεις των κειμένων για να μπορούμε να εργαστούμε εντός των προθεσμιών. Πριν από λίγους μήνες είχαμε ζητήσει να μάθουμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στις χώρες όπου ήδη ισχύει ο κανονισμός. Και δεν έλαβα καμία μελέτη το έργο λοιπόν αυτό έγινε, η έκθεση συντάχθηκε χωρίς την στήριξη της Επιτροπής μας. Θα έπρεπε λοιπόν οι υπάλληλοι μα να είναι λίγο πιο προσεκτικοί με τέτοιου είδου θέματα. Διότι δεν μπορεί στη διαδικασία τη συναπόφαση να έχουμε ακόμα την τεχνική και γλωσσική υποστήριξη που μα χρειάζεται και να μα λείπουν. Ε, να μα λείπει μάλλον η τεχνική και γλωσσική υποστήριξη που μα χρειάζεται. Ο κύριο Σούστα. Ευχαριστώ σύντομα, Πρόεδρε, γιατί το έχουμε ήδη συζητήσει. Όμως να θυμίσω ότι όσο υπάρχει συμφωνία επί τη ουσία μεταξύ του, του Κοινοβουλίου που έχει τοποθετηθεί με δύο ψηφίσματα και μία δήλωση και τη επιτροπή για τέτοια, τέτοια θέματα υπάρχει περίπτωση πρόοδου. Εδώ έχουμε κοινοτική, την κοινοτική μέθοδο που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Θα πρέπει λοιπόν από θεσμική άποψη να αξιοποιήσουμε την συμφωνία αυτή που υπάρχει και επιπλέον και με τα πολύτιμα στοιχεία που μα επισημαίνει η κυρία Μουσκαρντίνη βάσει και τη πρόταση τη Επιτροπή, από την οποία βεβαίω έχουν περάσει ήδη πέντε χρόνια. Οπότε προφανώ υπάρχει ανάγκη αναπροσαρμογή μα. Δεύτερη παρατήρηση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να καταγράψουμε την σύμπλευση των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτό το θέμα. Και στο Συμβούλιο, διότι αντιλαμβάνομαι ότι εντό Συμβουλίου τα εθνικά συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα είναι θεμητά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάντα ερμηνεύονται και από την άποψη της κάθε μιας χώρας ξεχωριστά. Σε αυτούς τους βιομηχανικούς όμως τομείς, εάν είχαμε την ίδια ευαισθησία που έχουμε για τα θέματα των τροφίμων λόγω χάρη, θα καταλαβαίναμε ότι δεν προσφέρουμε κάτι μόνον στην κατασκευαστική βιομηχανία της Ευρώπης, αλλά ιδίως στους πολίτες, διότι από τη μια υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή για την προέλευση των προϊόντων, τη σύνθεση, την θρεπτική τους ε, τις θρησκευτικές τους αξίες. Όμως όταν μιλάμε εδώ για τέτοιους τομείς, μιλάμε για φαντουργία, μιλάμε για κοσμήματα, μιλάμε για είδη οικοσκευής, όπως τα χαλιά ή τα ε, πρόσθετα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των δωματίων μας. Αφορούν και αυτά την υγεία και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Και, πολλές φορ... και εδώ δεν μιλάμε για παράξενα προϊόντα της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Μιλάμε για συγκεκριμένα είδη που επηρεάζουν το πώς κατασκευάζεται ένα, ένα, μια σκάλα, ένα αεροπλάνο ή το όταν φοράμε ένα ρούχο λόγου χάρη, παπούτσια. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώ είναι κατασκευασμένο το παπούτσι, το ρούχο που φοράμε. Το ίδιο εδώ και για τον καταναλωτή θα πρέπει να φροντίσουμε την προστασία του καθώ και την προστασία του βιομηχανικού τομέα που συζητούμε. Και θα πρέπει εδώ να ξεπεράσουμε τη διάκριση μεταξύ των υποστηρικτών των προμηθευτών και των υποστηρικτών της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο κανονισμό συγκλίνουν οι δύο αυτές διαφορετικές τάσεις. Θα πρέπει λοιπόν η προσέγγιση μα σε αυτόν τον κανονισμό να είναι επικοδομητική. Θα πρέπει να ασκήσουμε και την πολιτική μας επιρροή στα εθνικά μας κόμματα, στην κυβέρνησή μας, ώστε να φροντίσουμε στο Συμβούλιο να υπάρξει μια ευρεία συνένεση, γιατί εκεί θα είναι και το μεγάλο πρόσκομα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Um, e Ο κύριος Στέντι, ευχαριστώ. Συμφωνώ με όλα όσα είπε η κυρία Μουσκαρντίνη και τη συγχα... συγχαίρω για τα αγγλικά τη. Είναι πολύ καλύτερα από αυτά που οι δικοί μου συνεργάτε τα είχαν ετοιμάσει. Κύριε Σούστα, απλώ να πω κάτι. Πρόσφατα, πριν από έξι μήνε, αγόρασα ένα κουστούμι, πιστεύοντα ότι είναι ιταλική γραφή. Και ανακάλυψα ότι είχε κατασκευαστεί στο Χονγκ Κονγκ. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα με τι ετικέτε. Εντάξει, η ποιότητα καλή ήταν, αλλά είναι ένα πρόβλημα αυτό. Κατά τα άλλα, κυρία Μουσκαρντίνη, και απευθύνομαι και στου υπόλοιπου, η Επιτροπή Περιβάλλοντο μόλις προσφάτως ενέκρινε ένα κανονισμό για την ένδειξη προέλευσης στα τρόφιμα το κρέας και το καθεξής. Επέμενα για το θέμα αυτό επί χρόνια και νομίζω η ευκαιρία αυτή είναι τεράστια. Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά να τα δούμε από κοινού με την Επιτροπή σας. Διότι τώρα σε έναν τομέα έχουμε κάτι στα χέρια μας. Σα πάμε λοιπόν ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος όπως είπε και ο κύριο Σούστα, όταν έχει κανεί υπόψη ένα προϊόν το οποίο παράγεται και φτάνει στην τελική του μορφή στην Ευρώπη, αλλά έχει περάσει από διάφορες διαδικασίες, είναι δύσκολο να βάλουμε μία ετικέτα χώρας προέλευσης. Χώρας καταγωγής μάλλον. Αυτό δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία. Εκεί που έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας του προϊόντος, θα πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη. Βεβαίως αυτό θα ωφέλει μια ενταξη βεβαιως χώρες εισαγωγής. Κάποιε χώρε που εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν καλύτερη δουλειά. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ζήτημα εμπορικών φραγμών ούτε διάκριση. Εδώ μιλάμε για το πώ θα ωφεληθούν οι καταναλωτέ και οι πολίτε μα σε όλη την Ευρώπη. Είναι εξαιρετική λοιπόν η δική σα πορεία, όπω προδιαγράφετε, και να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε και τώρα λόγο στην Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω όσα ήδη υπόθηκαν. Συμφωνούμε ιδιαίτερως με την τελευταία παρατήρηση που έγινε. Ο κανονισμός αυτός σκοπό έχει να παράσχει πληροφορίες στους καταναλωτές, να τους ενημερώσει, ώστε να μπορούν να έχουν κάνει και αυτή μια υπεύθυνη επιλογή. Βεβαίως στο Συμβούλιο και αλλού υπάρχουν και φωνές που διαφωνούν και αναζητούμε εδώ την κατάλληλη ισορροπία στον κανονισμό αυτό μεταξύ των όσων θα ήθελαν ένδειξη της χώρας καταγωγής και όσων φοβούνται το κόστος που μπορεί να υπάρχει ιδίως ε, για την βιομηχανία μας και τους εμπορευομένους μας. Τώρα για το αν απαιτείται ειδική διαδικασία για την επιλογή των προϊόντων, τα στο παράρτημα, η δική μας πρόταση ήταν να υπάρχει μια διαδικασία επιτροπολογίας που θα επέτρεπε στο Ευρωκοινοβούλιο να έχει μια συνολική επισκόπηση του θέματος. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η μόνη δημοκρατική διαδικασία που μπορεί να προβλεφθεί με τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου είναι ακριβώς αυτή, οπότε θα υπάρχει και μεγαλύτερη διάρκεια για να γίνουν αλλαγές. Θα χρειάζεται μεγαλύτερος, περισσότερος χρόνος για να γίνουν αλλαγές στο παράρτημα. Όμως αυτό είναι στα δικά σας χέρια, εσείς θα αποφασίσετε εάν αυτό επιτυγχάνει την ε, σωστή ισορροπία μεταξύ της διάρκειας της διαδικασίας και τη δυνατότητα να τοποθετήσετε σε σχέση με τα προϊόντα που θα φέρονται ή θα προστιθείτε στο κατάλογο. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα από την πλευρά της Επιτροπής ε, το Κοινοβούλιο για την ε, συνεργασία και την επικοινωνία που είχαμε για το θέμα αυτό. Όπως και ο κύριος Σούστα, ελπίζουμε ότι αυτή η καλή ατμόσφαιρα συνεργασίας θα μεταφερθεί και στο Συμβούλιο Εκεί οι συζητήσει ήταν λιγότερο συνενετικέ, για να το πω έτσι. Ευχαριστώ. Uh, Ωραία. Κλείνουμε τη συζήτηση αυτή με την ε, εισηγήτρια, την κυρία Μουσκαρδίνη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που παρενέβησαν και τον συνάδελφο από την Επιτροπή. Νομίζω στο σημείο αυτό φαίνεται να υπάρχει ευρεία συμφωνία, η οποία μας επιτρέπει ακριβώ να έχουμε μια τελευταία συνάντηση και να καταλήξουμε σε τροπολογίες τον Ιούλιο, μετά να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τα τέλη Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Εδώ ανανεώνω την έκκλησή μου προς τους συναδέλφους. Εάν έχουν ειδικέ παρατηρήσεις να υποβάλουν ή αν έχουν τροπολογίες να υποβάλουν από κοινού, είμαι στη διάθεσή τους να τα συζητήσουμε μαζί. Επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Σούστα και τον κύριο Ρινάλντι οι οποίοι μαζί με μένα επεξεργάστηκαν τα θέματα αυτά, τα μελετήσαμε όλοι μαζί και από διαφορετικέ πολιτικέ οικογένειε υποβάλαμε κοινέ προτάσει. Νομίζω σε αυτή την επιτροπή ούτω ή άλλω όλοι έχουμε έναν τελικό στόχο. Να ε, εργαζόμαστε σκληρά σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχουμε αναλάβει. Διότι πολίτες ασχολούνται πολύ με το πώς οι